Ας αρχίσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Περιμένουμε μερικά λεπτά ε, για τον κύριο Βόσκι. Δυστυχώς, όπως θα μάθατε, ε, υπάρχει πένθος στην... Ε, Πολωνία. Ο διπλανός του Προέδρου μας, του Βογετσόφσκι, ο Μάρεκ Ρόζιακ, σκοτώθηκε σε μια επίθεση. Και επίσης και ένας άλλος βοηθός του κυρίου Βοζεβόσκι πληγώθηκε σοβαρά. Ως πρώτο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης θα σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ε, σε μνήμη του Μάρεκ Ρόζιακ. Παρακαλώ. Φυσικά, ε, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάρεκ Ρώσιακ και τις καλύτερες ευχές μας για ανάρρωση στον πληγωμένο βοηθό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί η σημερινή ημερήσια διάταξη. Ωραία, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις πριν από το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, ε, τα πρακτικά θα, θεωρούν, θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Ας ξεκινήσουμε με το σημείο 4. Ο ρόλος των γυναικών στην γεωργία και στην ύπεθρο. Ε, μετά από το ενδιαφέρον εργαστήριο για το ρόλο των γυναικών στην γεωργία, τον οποίο, όπως θα θυμάστε, οργάνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή μας. Ε, η κυρία Γέγκλε θα μας, παρα... θα μας παρουσιάσει την αρχική της ε, έκθεση. Πριν να της δώσω το λόγο, σας θυμίζω όλους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 16 Νοεμβρίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 16 Νοεμβρίου ώρα 12. Και τώρα με χαρά δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Ελίζαμπεθ Γέγκλε για να παρουσιάσει την έκθεση πρωτοβουλίας της. Ελίζαμπεθ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Ήδη ακούσαμε. Έχουμε χρόνο για την κατάθεση τροπολογιών καθένας από μας μπορεί λοιπόν να συμμετάσχει στις τροπολογίες και πιο πριν να έρθει σε επαφή και με τις ενώσεις γυναικών, γεωργών γυναικών και ενώσεις γεωργών να έρθει σε επαφή με όλους αυτούς. Αυτό ήδη στην πρώτη συζήτηση κατέστησα αφές ότι ήταν μεγάλο εγχείρημα. Στις 17 Νοεμβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργικής Πολιτικής που θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά θέματα. ο πρώτος πυλώνας, ο δεύτερος πυλώνας και ούτω καθεξής. Όμως με όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, το ζήτημα των γυναικών στην γεωργία και στον χώρο της υπαίθρου πολλές φορές στερείται κάλυψης και έτσι πολλές φορές πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των γεωργών στην Ήπεθρο και στη Γεωργία και είναι αυτό σαφές πλέον και, και για μένα κατέστη σαφές και το συνειδητοποίησα, επειδή όπως και οι περισσότεροι από εσά κατά κάποιο τρόπο, όπως και εσείς είχατε συμμετάσχει και έχω συμμε... Ε, μοιράσει την έκθεσή μου στις ενώσεις και συλλόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, που το προσχέδιό μου, το προσχέδιό μου αυτό μπόρεσαν να το διαβάσουν και μπόρεσαν να εξοικειωθούν. Και Ό,τι υπέβαλαν ως προτάσεις ε, από την πλευρά τους ε, και από συναδέφους αφετέρου, αλλά και από ενώσεις ε, και άλλους, για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό στοιχείο. Για αυτή την πρώτη μορφή του προσχεδίου μου, με όλα αυτά τα οποία κατατέθηκαν, ξαναέγραψα την έκθεσή μου και αυτή είναι τώρα η μορφή, το η έκθεσή μου που έχετε στα χέρια σας. Τις προηγούμενες δεκαετίες η ΚΑΠ η κοινή αγροτική πολιτική βασιζόταν στην θετική οικονομική εξέλιξη των της γεωργίας και προς αυτήν στόχευε. Μελλοντικά όλο και περισσότερο θα πρέπει να διαμορφώνουμε ικανούς ε, για ανταγωνισμό και παραγωγή νέους χώρους και θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις προσπάθειες. Μέσα σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου δράσης είναι ανάγκη να λάβουμε υπόψη το πιστεύω ακράδαντα, τις ανάγκες αλλά και το δυναμικό των γυναικών στους χώρους της Υπέθρου. και να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Η πείρα δείχνει, η οικονομία το δείχνει και όλες οι παρεμβάσεις το καταδεικνύουν ότι η ποιότητα διαβίωσης και κυρίως η αποτελεσματικότητα στην Ήπεθρο εξαρτάται από την παρουσία των γυναικών και από την πολύμορφη συμμετοχή των γυναικών στις δράσεις αυτές. Έχουμε πολλές φορές ε, τις περιπτώσεις ε, περιοχών που εγκαταλείπονται από γυναίκες και νέες γυναίκες και έτσι δεν θα έχουν καμιά πρόπτικη να επιβιώσουν στο μέλλον αυτοί οι χώροι και καταδείχθηκε ότι με την υποστήριξη των γυναικών και για σημαντικά τέτοια εγχειρήματα για την κοινωνία που υποστηρίζονται από αυτή τη δράση και αυτό πάλι ήταν ένα μήνυμα το οποίο μας δόθηκε με κάθε σαφήνεια. Και στη γεωργία την ίδια ο ρόλος της γυναίκας είναι ουσιοδέστατος. Έχουμε γυναίκες που κατά το παρελθόν συνεισέφεραν για την προσαρμογή ακριβώς ε, όπως ήταν αναγκαίο της γεωργίας. Η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας ακόμα περισσότερο πήρε σάρκα και οστά και εξειδικεύτηκε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπόρεσαν καινοτόμε προσφορές να τις αποδεχτούν και να συμμετάσχουν έτσι και πολύ με αυτό το ζήλο των γυναικών μπόρεσαν να προχωρήσουν θετικά. Μια σημαντική άλλη ήταν η ενδυνάμωση των γυναικών μέσα στο πλαίσιο των ενώσεων, των συλλόγων, συνεταιρισμών και οργανώσεων. Αυτό απορρέει από το αίτημα για μια ποσόστοση παρουσίας των γυναικών στις ενώσεις και συλλόγους που όπως γενικότερα εντάσσεται αυτή η διατύπωση στην έκθεσή μου απαιτεί μια επαρκή και κατάλληλη, κατάλληλα προσαρμοσμένη παρουσία και εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτά τα όργανα. Καθώς επίσης ε, οι γυναίκες στην γεωργία όπως είναι εξακολουθεί και είναι ένα μεγάλο θέμα και ζήτημα το οποίο θα εκπονήσουμε και θα αναλύσουμε Χαίρομαι για τις τροπολογίες, προσδοκώ αδειμονώ να τις δω. Με τις τροπολογίες θα έρθω σε επαφή με όλους τους συναδέλφους που θα έχουν καταθέσει αυτές τις προτάσεις για να, να δούμε αυτά τα πράγματα, να ε, τις εξετάσω και να έχουμε μια καλή έκθεση στο τέλος ε, που θα ανταποκρίνεται στη συζήτηση και στο περιεχόμενο της συζήτησης για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής προς όφελος των γυναικών στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ελίζαμπεθ. Ας ανοίξουμε αμέσως τη συζήτηση. Ο κύριος Τζασάλα ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαιρετικό το έγγραφο αυτό για το ρόλο των γυναικών στη γεωργία και την ύπεθρο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και την περασμένη εβδομάδα έμαθα και εγώ πόσες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί στη Δυτική Πολωνία πήραν μέρος σε κοινωνικές διαβουλεύσεις εκατοντάδες άνθρωποι εξών και γεωργοί από την Ήπεθρο σε εγκαταστάσεις ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και έμαθα ότι οι γυναίκες που πήγαιναν εκεί δήλωναν ότι χρειαζόντουσαν ηγέτιδες για να οθηθούν έτσι διάφορα προγράμματα. Πρέπει να οθήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ήπεθρο και ιδίως την ηλεκτρονική επιχείρηση οι γυναίκες πρέπει να δημιουργήσουν ιστοσελίδες και να μπορούν να λειτουργούν ηλεκτρονικά μαγαζιά στην Ήπεθρο, διότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές και καταναλώτριες επιζητούν βιολογικά ρόφημα. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες όπως ε, παιδική σταθμή στην Ήπεθρο χρειάζονται απολύτως γιατί η ύπαρξη τέτοιων παιδικών σταθμών βοηθά τις γυναίκες να παραμείνουν στην ύπεθρο. Επίσης τις βοηθάει και αργότερα να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Διότι κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου μαθαίνουν τα παιδιά και του παιδικού σταθμού τα βασικά στοιχεία και πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε και τις οργανώσεις των γυναικών στην Ήπεθρο που είναι τόσο σημαντικές για την πολιτιστική εξέλιξη των περιοχών αυτών στην Πολωνία. Υπάρχουν οργανώσεις αγροτισών που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Είναι και οι μεγαλύτερες του είδους του στη χώρα. 260 στην περιφέρειά μου και μόνο υπάρχουν και συνεισφέρουν πολύ θετικά στη λειτουργία διαφόρων ε, ε, πολιτιστικών και άλλων προγραμμάτων. Οι γυναίκες που πήγαν στις συνεδριάσεις αυτές τόνισαν ότι χρειάζονται ανταλλαγές βελτίστων πρακτικών συζητήσεις για να μπορέσουν να συμβάλλουν και αυτές στην κατάστροφη της στρατηγικής μίας ανάπτυξης της υπαίθρου. Συγχαίρω εκ νέου την εισηγήτρια. Έχω ορισμένες τροπολογίες βέβαια που αφορούν ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, ιδίω την ηλεκτρονική επιχείρηση, καθώς και την πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και τη στήριξη των γυναικείων οργανώσεων στην Ήπεθρο. Στο. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Γέγκλε για την πάρα πολύ ευρεία έκθεση, πάρα πολλά θέματα συμπεριέλαβε από αυτά που συζητήσαμε και την ευχαριστώ γι' αυτό. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα επειδή μιλάει για το ρόλο των γυναικών στην πολυλειτουργικότητα της Γερμανίας. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο που έχουμε χρόνο να έχουμε ανατροφοδότηση από τις γυναικείες οργανώσεις γιατί αυτό σημαίνει ότι προσπάθειά μας εμπεριέχει μεγαλύτερη συνεργασία και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πολίτες μας στις εκθέσεις που γράφουμε εδώ και να ξέρουμε ότι κάπως συμμετέχουν κι αυτοί, κάποιο λιθαράκι βάζουν κι αυτοί. Ένα-δυο σχόλια και ένα-δυο ερωτήσει για τον εισηγητή. Νιώθω ότι... Ε, είναι σημείο κλειδί η θέση των γυναικών ε, στην γεωργία και πρέπει να δούμε πώς θα συμμετέχουν και να αναπτύξουμε το δυναμικό τους. Μου αρέσει ιδιαίτερα η παράγραφος 17 όπου μιλάμε για τις γυναίκες επιχειρηματίες και στο πλαίσιο της καινοτομίας ε, είναι πολύ σημαντικό ε, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 να περάσουν και στις γυναίκες στη Γεωργία Υπήρχε ένα αρχικό σχέδιο κειμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το οποίο η Γεωργία θα παίξει πολύ μικρό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι κάθε συγκυρία έμφασης του ρόλου της Γεωργίας είναι ευπρόσδεκτη. Πράγματι μπορεί να συμβάλλει η Γεωργία στην επιτέξη των στόχων για το 2020 και ο ρόλος των γυναικών σε αυτό επίσης είναι κάτι σημαντικό για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και πάλι έχει σημασία να στοχεύσουμε σε αυτά ε, υπάρχει και το ηλεκτρονικό επιχειρήν και αυτό είναι σημαντικό και αυτό να το βάλουμε μέσα. Μια-δυο ερωτήσεις για την εισηγήτρια παρακαλώ. Στην παράγραφο 6 καλείται για προϋποθέσεις πλαισίου για την Ήπεθρο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με το πλαίσιο, με τις προϋποθέσεις πλαισίου, framework conditions, επίσης η παράγραφος 1 ε, ε, επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής ενοποίησης η υποστήριξη των γυναικών. Και πάλι δεν βλέπω πολύ καλά ποια σχέση έχουν. Ίσως η εισηγήτρια μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα. Στην παράγραφο 4 επίσης, παρόλο που συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Δεν ξέρω πώς η μέρημνα για τους ηλικιωμένου και το παιδί συνδυάζεται. Περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις της κυρίας Γέγκλη και την ευχαριστώ για άλλη μια για τη δουλειά της. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν. <clears throat> <clears throat> Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Γέγκλε για την έκθεση εμπεριέχει πάρα πολλά που απερίφραστα τα σημεριζόμαστε χωρίς επιφυλάξεις. Το ότι πρέπει να συνδυαστεί με τη μεταρρύθμιση στην πολιτική γεωργίας πρέπει να καταστεί σαφές. Αναφέρεται ένα κύριο πρόβλημα ότι πολλές προσοντούχες γυναίκες εγκαταλείπουν το χώρο της υπαίθρου επειδή δεν έχουν δυνατότητα να επιβιώσουν από το εισόδημά τους και στην γεωργία κυρίως ε, και πρέπει να είναι τα εισοδήματα επαρκή στην, από τη γεωργία για να παραμένουν οι γυναίκες ε, στην υπαίθρο. Μια πολύ σημαντική πτυχή που νομίζω λίγο περισσότερο θα έπρεπε να τονιστεί είναι η δυνατότητα για γυναίκες ε, να περιθάλπουν ε, όπως και συμβαίνει και στο χώρο των πόλεων και τα παιδιά τους, να φροντίζουν τα παιδιά τους. Αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται για τις γυναίκες τόσες θέσεις να υπάρχουν για την μέρημνα των παιδιών. Υπάρχει όμως έλλειψη εκεί και πρέπει να επεκταθεί η δυνατότητα φροντίδας των παιδιών. Για το σημείο 20 που λέτε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς σε πολλούς φορείς και όργανα όπου πριν τα ανέβουν οι άντρε, για να το πω ιδιαίτερα επιφυλακτικά στη διατύπωσή μου, θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να διαμορφωθεί, να διατυπωθεί αυτό το σημείο. Υπάρχουν πολλέ συζητήσει με ιδέε πώ μπορεί αυτό να βελτιωθεί και με ποσοστώσει που μπορούν να εισαχθούν. Γιατί κατά τα άλλα, αν δεν είμαστε εξειδικευμένοι, είναι μια έκκληση που την ξεχνάει κανεί πολύ συχνά αμέσω μετά. Και σε αυτό το σημείο ίσως θα έπρεπε να επικεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας και στο ότι οι γυναίκες ως ανεξάρτητες επιχειρηματίες στη Γεωργία καλό είναι να προσφέρονται προσόντα ώστε οι γυναίκες να μπορούν να αναλάβουν νέες εκμεταλλεύσεις και να στήσουν μια νέα ζωή, ε, να μπορούν να στηρίξουν τη ζωή τους στον τομέα της υπαίθρου από αυτή τη δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Ο Αντιπρόεδρος Πόλτσο την... έχει το λόγο. Eh, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Γέγκλε. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση η έκθεση που έχετε υποβάλει κυρία Γέγκλε και πρέπει να πω ότι εγώ πραγματικά αυτή τη φορά δεν μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Χάκιν. παρόλα αυτά πρόκειται για το ότι η Γεωργία θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω στην εξέτασή της από μας από την παραγωγή κάποιων γεωργικών προϊόντων. Η ζωή λοιπόν στην Ήπεθρο είναι μια σύνθεση από διαφορετικές πολυσχηδείς δραστηριότητες. Υπάρχουν διάφορες πηγές εισοδήματος στην Ήπεθρο. Εδώ όμως πρόκειται μεταξύ άλλων και για την φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Και αυτό είναι σημαντικό για να έχουν οι γυναίκες την δυνατότητα να αποφασίζουν ελεύθερα για τη ζωή τους και τη δραστηριότητά τους και το χρόνο τους. Και είναι σημαντικό σε αυτό να δημιουργηθούν και θέσεις απασχολήσεις για γυναίκες. Θα ήθελα εδώ μόνο μία μικρή παρατήρηση να κάνω. Ίσως κάπου κάπως προκλητικού χαρακτήρα αν θέλετε για να προκαλέσω μια αντίδραση. Αυτό που θα ήθελα είναι να δούμε στο 19 στην ε, όχι, είναι η 18. Στο 18 λοιπόν της έκθεσής σας τι λέγεται, ότι οι γυναίκες λέει στη Γεωργία συχνά είχαν υψηλό ποσοστό αναφέρεται σε κάθε Καθένας μπορεί να μάθει βέβαια ε, το επάγγελμα που επιθυμεί. Προφανώς όμως ένα μέρος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενισχυμένα βασιζόταν στο εργατικό δυναμικό των γυναικών. Υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με τη γεωργία όχι μόνο στη δική τους εκμετάλλευση, αυτές βέβαια έχουν και μια ιδιωτική ζωή και που μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται σε σχέση με εκείνες τις γυναίκες που έχουν παντρευτεί άντρες γεωργούς σε σχέση και με το πώς οι άντρες γεωργοί διαμορφώνουν τη ζωή τους. Θα έλεγα όμως ότι η έκθεση πέρα από αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Τόσο καλή που θα την υπερψηφίσω χωρίς να διστάσω. Και σε αυτό το σημείο θα καταθέσω αίτηση τροπολογίας, μια τροπολογία. Η έκθεση κατά τα άλλα είναι πλήρης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πόλσεν. James Nicholson. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πάλι και συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. Είναι πολύ καλή η έκθεση. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που διατυπώθηκαν ήδη και νομίζω ότι κάτι που πρέπει να αποδεχθούμε, ανεξάρτητα από το που ζούμε, ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές, η Ήπεθρος γενικά, τα τελευταία 30-40 χρόνια βαθμιαία άλλαξαν και αυτή η αλλαγή προκλήθηκε με βάση διαφορετικές ανάγκες και διάφορα κριτήρια και διάφορες προκλήσεις. Κάπου οι γυναίκες ε, έφυγαν και αναζήτησαν αλλού εργασία και αυτό δημιούργησε και προβλήματα στη γεωργική οικογένεια. Αλλά και επειδή δεν υπάρχουν ε, ρόλοι και επαγγέλματα να αναλάβει η γυναίκα στις ε, γεωργικές περιοχές, υπάρχει αυτή η φυγή. Ε, και δεν χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στην Ήπεθρο, τα τεχνολογικά εργαλεία. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι η κατάρτιση. Ε, μια από τις αδυναμίες της γεωργίας είναι ότι πολλοί γεωργοί είναι τόσο πολύ άσχαλοι φροντίζοντας τα ζώα τους και όλα τα άλλα που ξεχνούν την πλευρά της τεχνολογίας. Και πρέπει, χρειάζονται κατάρτιση για να ανταποκριθούν στις καινούριες προκλήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε εκεί να επιτύχουμε μεγάλες βελτιώσεις. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις μετά το 2013 και είναι πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο εταίροι, συνεταίροι, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτριες γεωργικών εκμεταλλεύσεων πλέον. Υπάρχουν πάρα πολλέ που έχουν ορνηθοτροφία ή χειροστάσια. Δεν είναι καθόλου αδύνατο ή ασύλληπτο αυτό. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνει. Και φυσικά αναπτύσσεται η κοινωνία, μεταβάλλεται, οι γυναίκες μπορούν να φέρουν και καινούργιες ιδέες ο τουρισμός, εργασίες, τις εκμεταλλεύσεις, η, η ανάπτυξη νέων ιδεών για την αγροτική οικονομία, για τη γεωργική οικονομία, Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε όλοι να επιτύχουμε είναι καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους όσους ζουν στις γεωργικές περιοχές. Και βεβαίως πράγματι πρέπει να αναπτυχθούν και οι δομές φροντίδας του παιδιού στις αγροτικές περιοχές. Κάμπολας Αγκόστο, Λουίς, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ε, επενώντας την εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και από πλευρά σα κοιόδου ε, εισηγήτρια τη Σοσιαλιστική Ομάδα που σήμερα δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί και μου ζήτησε να διαβιβάσω τη σύμφωνη γνώμη τη με το γενικό πλαίσιο ε, τοποθέτηση τη έκθεση έκθεσης ενώπιον του προβλήματος. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι οι πολιτικέ που ακολουθούνται πάντα. Είναι πίσω από έναν μεγάλο πολιτικό βρίσκονται γυναίκες. Μια μεγάλη γυναίκα. Εδώ ιδιαίτερα για την ε, γυναίκα που βρίσκεται πίσω από κάθε γεωργό. Είναι μεγάλες αυτές οι γυναίκες. παρόλα τις δυσκολίες ε, της γεωργικής ζωής ε, ασκούν όλες τις δραστηριότητες ε, που δεν ασκούν κανονικά οι άνδρες γεωργοί και κυρίως σε μια χρονική στιγμή όπου οδηγούμαστε σε μια συμπληρωματικές δραστηριότητες όσον αφορά την γεωργική πραγματικότητα. Όταν κάνουμε λόγο για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων κυρίως είναι αυτές οι δραστηριότητες ε, που ασκούνται από γυναίκες και που διευθύνουν οι ίδιες οι γυναίκες. Όταν οι ίδιες αυτές οι γυναίκες είναι επικεφαλής εκμεταλλεύσεων γεωργικών. Γι' αυτό ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να εξισώσουμε το καθεστώς τους και να τους δώσουμε ένα ρόλο σημαντικό που πρέπει να τους αρκεί τότε κάνουμε αυτό που πρέπει για τη γεωργία και το χώρο της υπαίθρου. Και αυτό είναι ο τελικός στόχος τελικά και της κυρίας Γέγκλε. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας και εξ ονόματος της Σκιώδους εισηγήτριάς μας και εξ ονόματος της πτέρυγάς μας ότι δεσμευόμαστε και η τελική έκθεση θέλουμε ακόμα να είναι καλύτερη αν είναι δυνατόν και έτσι την δεχόμαστε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ Λουίς. Ο κύριος Καλνιέτε. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu teikt, ka man bija iespēja iepazīstināt. Ευχαριστώ. Είχα τη δυνατότητα να διαβάσω την έκθεση και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι αφού τη διάβασα την έκθεση Άκουσα από γυναικείες οργανώσεις στη Λιθουανία ότι αυτά ακριβώς ήθελαν να ακούσουν. Τονίζει ιδιαίτερα πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συνεισφέρουν στην οικονομία δημιουργώντας ένα δίκτυο επιχειρηματιών γυναικών στην Ήπεθρο. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η προσπάθεια διευκόλυνσης με χρηματική στήριξη των ε, οργανώσεων γυναικών. Είναι σημαντικό νομίζω να τις προσέξουμε τις οργανώσεις αυτές και τη συνεργασία που μπορούν να προσφέρουν για να μπορούν οι γυναίκες πιο εύκολα να αρχίσουν μία επιχείρηση έμπειρες γυναίκες θα μπορούν έτσι να χρησιμεύσουν στις ε, νεότερες για συμβουλές. Θα ήθελα λοιπόν ακόμη μια φορά να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κλείνω τη συζήτηση. Ο Αντιπρόεδρος Μποβέ. Έχετε το λόγο. Oui, euh, de la même manière, euh, je... Κοιτάξτε, και εγώ, και εγώ υποστηρίζω την έκθεση είναι ενδιαφέρουσα και αναφέρει πάρα πολλά στοιχεία. Μερικά από αυτά θέλω να αναφέρω. Ένα, σε σχέση με την ψηφοφορία που κάναμε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα για την μητρική άδεια, θα έπρεπε ίσως να βάλουμε και αυτό το σημείο εδώ, ένα σημείο για τη μητρική άδεια που πρέπει να διαθέτουν, που πρέπει να έχουν οι αγρότησες για να αυξάνεται και για αυτές είναι νομισμένη μητρική άδεια. Και δεύτερον, κάτι που σχετίζεται με διάφορα σημεία του σκεπτικού της επεξηγηματικής έκθεσης, η αναγκαιότητα να τα συνδέσουμε αυτά και με τη συζήτηση για την ΚΑΠ όπως αναφέρει το προσχέδιο έκθεσης που λάβαμε, να επιμείνουμε στα μικρά αγροκτήματα όπως κάνει η Κομισιόν γιατί είναι σημαντικό η έννοια της συνεκμετάλλευσης που υπάρχει σε ορισμένες χώρες να αναγνωριστεί να υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών και μεταξύ των αγροτών γιατί σε μερικές χώρες η νομοθεσία δεν προβλέπει ισότητα και εδώ πρέπει να γίνει μια εναρμόνιση για την αναγνώριση αγροτών και αγροτισών επίσης όρισης. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Και πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Γέγκελ, έχουμε την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον κύριο Μπρόζη έχουμε σήμερα μαζί μας. Παρακαλώ. Um, Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Γέγκλε για την πρωτοβουλία αυτή. Φυσικά δεχόμαστε πολύ θερμά αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσω του δεύτερου πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής τη δυνατότητα να στηρίξουμε τις γυναίκες. Η κυρία Γέγκλε ε, μιλά για Eigen Dynamics, για ίδια δυναμική, ε, για επιχειρηματικές δράσεις ε, ίδιες, οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν χρηματοδότησης από τα προγράμματα πρωτοβουλίων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη, για τη χάραξη της ε, μελλοντικής πολιτικής. Για τις γυναίκες σας στη Γεωργία θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη έχουν λάβει τώρα τη νέα οδηγία για την υλοποίηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και στα πλαίσια των αυτοαπασχολούμενων. Ελπίζουμε ότι οι σύζυγοι των γεωργών επιτέλους θα τύχουν τις προσοχής που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρόζε. Και τώρα η Ελίζαμπε έχει τον λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις και να καταλήξει. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους, γυναίκες και άνδρες. Και αν επιτρέπετε να ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρηση ακριβώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα και αυτό που είπατε είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, ακριβώς μέσα στο νέο πλαίσιο της συζήτηση για τη νέα αγροτική πολιτική, αυτά τα οποία σε αυτή την έκθεση που είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας προτίθενται, σε τμήματα και μέρη να αντανακλώνται από αυτή τη νέα πολιτική. Αυτή είναι η επιθυμία μου και αυτή είναι η επιθυμία μας. Αυτό είναι η εξήγηση, το σκηνικό αυτής της έκθεσης και των στοιχείων της. Γι' αυτό ας προσπαθήσω κάπως να αναφερθώ και να ανταποκριθώ στους συναδέφους. Προσφέρω σε όλες τις συναδέφους και όλους τους συναδέφους την δυνατότητα κατηδίαν να έρθουμε σε επαφή, να συζητήσουμε και να δούμε τις προτάσεις αυτές. Έχουμε αρκετό, πολύ χρόνο και θέλω να το πω και αυτό. Θα ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου 2011 στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και τον Μάρτιο του 2011 θα περάσουμε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Έτσι υπάρχει χρόνος στα κράτη μας να έρθουμε σε επαφή με ενώσεις και συλλόγους γεωργών να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θέλω ευρύτατη δημοσιότητα, δημοσιότητα να διασφαλιστεί για αυτό το θέμα και τα στοιχεία του. Τώρα, επί της ουσίας, ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα θέματα στα όσα μου είχατε πει αναφέρονται και εν και με τα ίδια αιτήματα τα οποία διατυπώνονται τώρα που κατά κάποιο τρόπο αποδυνάμωσα στην έκθεσή μου εγώ. Και πρέπει να ξέρει κανείς ότι μια τέτοια έκθεση έχει συγκεκριμένο περιορισμένο αριθμό ψηφίων που πρέπει να εμπεριέχει. Και γι' αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση να δω αν μπορούμε με τροπολογίες να καλύψουμε κάποια αιτήματα. Περίθαλψη και φροντίδα παιδιών και ατόμων από γυναίκες στην Ήπεθρο, όπως και το ακούσαμε και για, από την Ιταλία, κάτι το οποίο για μας στη Γερμανία ήταν ε, άγνωστο. Νομίζω ότι και για το μέλλον είναι μια πολύ καλή ιδέα. Το θέμα είναι πώς κάτι τέτοιο μπορούμε να το προτείνουμε και να το εντάξουμε σε αυτό όσον αφορά την υποστήριξη και συμμετοχή σε αυτές τις θέσεις και από πλευράς του συναδέρφου αναφέρθηκαν τα στοιχεία αυτά, πρέπει να δοθεί συνέχεια. Γυναίκες ως ε, επιχειρηματίες και γυναίκες ο ρόλος των γυναικών να ενδυναμωθεί κυρία Χάρκιν. Σε αυτά τα οποία η κυρία Πάουλσεν είπε και κατέστησε σαφή είναι και αυτά για μένα πολύ σημαντικά. Κυρία Πόλσον, αν επιτρέπετε να απαντήσω στην ερώτησή σας, πιθανώς αυτό το οποίο βλέπετε εσείς ως πρόβλημα είναι γλωσσικό πρόβλημα. Εγώ στην Γερμανία, στον χώρο της Υπέθρου, από πλευράς της γλώσσας, και με γυναίκες και εργαζόμενους στην, ε, συνεργάτες στην οικογένεια άλλοι ζουν στην πόλη άλλοι ζουν στον στο χώρο της Υπέθρου. γλωσσικά το διατύπωσα αυτό με έναν όρο που διαφοροποιεί τα πράγματα. Μπορεί να είναι επιχειρηματίες γυναίκες, αλλά εγώ αναφέρθηκα στο ότι οι γυναίκες που ζουν εκεί κάπως γλωσσικά πρέπει να το δούμε και είναι σαφές ότι αυτό ίσως δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αυτό που θέλω να δημιουργείται με σαφή εντύπωση είναι οι γυναίκες στο χώρο της υπαίθρου να μπορούν να είναι ε, ανεξάρτητες επιχειρηματίες. Μπορούν όμως να είναι μέλη της οικογένειας ε, συνεργαζόμενοι σε μια οικογενειακή εκμετάλλευση παράδειγμα. Επίσης γυναίκες που στον χώρο της υπαίθρου ζουν και ασκούν ένα επάγγελμα ως μισθωτές κάπου. Και αυτό πρέπει να δούμε. Να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης εργασίας των γυναικών στην Ήπεθρο και έτσι. Ή και ως γυναίκες επιχειρηματίες ξεχωριστά, ανεξάρτητες να μπορούν να υπάρχουν στο χώρο της υπαίθρου, όπως αναφέρουμε. Το θέμα της φροντίδας παιδιών, το έχω απαντήσει και με αυτή την προσέγγιση. Εξεπλάγει ιδιαίτερα με πόσο έντονο τρόπο μου τέθηκε αυτό το θέμα και σήμερα πάλι το θίξατε. Ζητεί, απαιτεί συνθήκες πλαίσιο να διασφαλιστούν. Είναι το σημείο 6 κυρία Χάκιν. Έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις ε, όσον αφορά την ε, δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τις παρατηρήσεις σε σχέση με τη δική μου έκθεση. Ως συντάκτρια μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Όμως υπάρχουν και διαφορετικές πηγές διασφάλισης εισοδήματος. Και όταν κάνουμε λόγο για μια κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να σκεφτούμε τι μας αφορά εμάς, αλλά εσείς όλοι είσαστε και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε αυτά τα αιτήματα και να τα εντάξουμε. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση όπως την υιοθέτησα. Μετά και για τη στοχοθέτηση και τους προσανατολισμούς συνάδελφε κάτι πολύ χρήσιμο τι ωφελούν όλα μας τα προγράμματα αν παραμείνουν αποψηλωμένα αποψηλωμένη από α, ανθρώπους και κατοίκους θα έχουμε ακόμα πιο πολλές δυσκολίες άρα πρέπει πρόληψη να ισχύσει προληπτική αντιμετώπιση και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των ανθρώπων στην ύπεθρο αναμένω τις τροπολογίες σας όμως εισαγωγικά ήδη το είχα προαναφέρει ότι ζητήθηκε ποσόστοση, ποσόστοση μέχρι 40%, 40% ή τουλάχιστον αυτή ήταν μια πρόταση, όμως επέλεξα τον όρο ενδεδειγμένη εκπροσώπηση, σκόπιμη κατάλληλη εκπροσώπηση των γυναικών που πρέπει να διασφαλίζεται. Σε αυτό το σημείο θέλω ένα πράγμα να καταστήσω σαφές και ανήκει και το επόμενο σημείο σε αυτό. Προσόντα, προσοντούχες γυναίκες στη γεωργία, σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Εξειδικευμένα πράγματα πρέπει να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία που θέλω να ενθαρρύνω τις γυναίκες και ενώσεις ε, αυτό το οποίο είναι εφικτό και δυνατό να το κάνουν προσωπικά για αυτή την, για την ευόδοση αυτού του στόχου. Παρακαλώ στις συζητήσεις με τις ε, χώρες σας να το αναφέρετε αυτό. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Πολλά μπορούν να γίνουν από τις γυναίκες ήδη σήμερα. Καμιά φορά πρέπει ας το πω αυτό να δοθεί μια όθηση σε αυτές ε, να το πω στα σουηβικά της Σουηβίας ε, της επαρχίας μου να δώσουμε μια βοήθεια, ένα χεράκι, μια όθηση να γίνει αυτό. Πολύ σωστά το είπατε. Στα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες πολλά πράγματα σε τεράστιο βαθμό άλλαξαν στους χώρους της υπαίθρου. Χαίρομαι λοιπόν και προσδοκώ τις τροπολογίες. Και έτσι σε σχέση με αυτές τις αλλαγές πρέπει να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας και να οδηγηθούμε σε μια βελτίωση της διαβίωσης για όλους. Αυτό είναι η διατύπωση που επελέγει. Τώρα, αν θα εντάξουμε την άδεια μητρότητα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την έκθεση, να δούμε και νομικά αν μπορεί να γίνει, μέσω μια τροπολογίας ίσως. Αλλά ομολογώ, εγώ ομολογώ, ότι στο τέλος είπα όχι, να μην το εντάξω στην έκθεσή μου, υπό το δικό μου πρίσμα, γιατί είναι ένα θέμα που ανήκει στην επικουρικότητα στο θέμα των κρατών μελών. Είναι η προσωπική μου άποψη που εκφράζω εγώ εδώ. Είμαι όμως πρόθυμη αν υπάρξουν κάποιες προτάσεις να τις δω, να δω αν μπορώ να τις δεχτώ και να τις εντάξω. Κύριε Μποβέ, εσείς τι είπατε, είπατε δημιουργήσατε τη διασύνδεση στην ΚΑΠ κάνοντας λόγο για κοινέ εκμεταλλεύσεις, ε, κοινέ επιχειρήσεις και σε σχέση με άνδρες και γυναίκες ε, πώς αυτό διαμορφώνεται. Και στην ΚΟΠΑ και άλλες οργανώσεις ε, έκανα αυτή τη συζήτηση. Αδειμονώ να δω ποιες θα είναι οι τροπολογίες που θα έχω. Και σε σχέση με τα κράτη-μέλη τι θα πούν σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα είναι δεδομένο, το ξέρω. Η εφαρμογή όμως νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η υλοποίηση και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Προσδοκώ να δω τις τροπολογίες και να έχω και τις συζητήσεις που θα πρέπει να έχουμε για να μην έχουμε εκατοντάδες τροπολογίες που θα ψηφίσουμε στο τέλος αλλά να συναντηθούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις τροπολογίες, ποιοι συμβιβασμοί μπορούν να επιτευχθούν για να έχουμε ένα καλό κείμενο στο τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ελίζαμπεθ Γέγκλε, πολύ καλή δουλειά. Υπενθυμίζω και πάλι σε όλους τους συναδέλφους ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών για την έκθεση Γέγκελ είναι 12 η ώρα στις 16 ε, Νοεμβρίου. Ας περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, γεωργία και διεθνές εμπόριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως το ξέρετε, οι διεθνείς συμφωνίες για το εμπόριο και η απελευθέρωση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων έχουν τεράστιες επιπτώσεις για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, να εγγυηθούμε ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, ε, της ορθής μεταχείρισης των ζώων, της υγιεινής των τροφίμπων δεν πρέπει να τροποποιηθούν από μια αγορά ανίκανη να αναγνωρίσει τις κοινωνικές αξίες που ενσωματώνει το προϊόν. Στο προϊόν πρέπει να απαλείψουμε τις τρευλωτικές επιπτώσεις και θα πρέπει οι διεθνείς παίκτες ε, ε, να μπορέσουμε μάλλον τις υποχρεώσεις, ε, τις, τις υποχρεωτικές διατάξεις τις οποίες εφαρμόζουμε να τις μετατρέψουμε σε μεγάλα πλεονεκτήματα για μας. Ε, τα κοινωνικοπεριβαλλοντικά πρότυπα πρέπει και αυτά να τα μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Ο κύριος Παπαστάμκος είναι ο εισηγητής αυτής της έκθεσης. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι ε, επίσης συναφή επιτροπή υπό την έννοια του άρθρου 50 του κανονισμού. Τον λόγο έχει ο κύριος Παπαστάμκο και σας θυμίζω αμέσως ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 10η Νοεμβρίου. Γιώργο, έχει τον λόγο. Ε, θα αναφερθώ σε μερικές μόνο πτυχές ε, της έκθεσης και της ε, πρότασης ψηφίσματος τις οποίες έχετε αναχείρα σας. Ε, σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής, θεωρώ ότι η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής καθίσταται άκρο σημαντική. Στο πλαίσιο της ε, εξωτερικής εμπορικής πολιτικής, η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζεται να διασφαλίζει τον πολιτουργικό ρόλο της γεωργίας, όπως τον βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό μοντέλο. Η διαπραγματευτική προσέγγιση της Κομισιόν, η οποία προβαίνει σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας, έναντι αυξημένης πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών στους τομείς των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών ε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και κατά τη γνώμη μου δεν είναι αποδεκτή. Η Κομισιόν θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολογήσεις του αντικτύπου στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, οι οποίες να δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και να επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες θέσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις. Ε, παραδείγματι, κατά τη γνώμη μου, είναι επικριτέα η απόφαση της Κομισιόν για επανέναξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της Μερκοσούρ. Δεν λέω αν θα πρέπει να έχουμε σχέσεις και είμαι υπέρ των σχέσεων με τις χώρες της Μερκοσούρ, αλλά αναφέρομαι στην τακτική ε, συστάση της Κομισιόν. Είναι επομένω επικριτέα η απόφασή της για επανέναξη των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της Μερκοσούρ χωρίς να προηγηθεί λεπτομερής εκτίμηση του αντικτύπου στον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Δεδομένου ότι διεξάγεται παράλληλα πληθώρα εμπορικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να υιοθετηθεί για κάθε επιμέρους γεωργικό τομέα της Ένωσης μία προσέγγιση, μια τέτοια προσέγγιση που θα διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών καθώς και τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος και των γεωργικών αγορών στην ε, ε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αφερθώ σε ένα μόνο παράδειγμα. Οι παραχωρήσεις που ανέλαβε η Κομισιόν στον τομέα της ζάχαρης έναντι χωρών της Λατινικής Αμερικής θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Ταμέα Ζάχαρης, ο οποίος υπέστη, ως γνωστόν, ήδη σοβαρές επιπτώσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αγοράς ζάχαρης το 2006 η Κομισιόν συχνά προκρίνει ως λύση τη χρηματική αποζημίωση έναντι των αρνητικών επιπτώσεων από το άνοιγμα της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζω ωστόσο ότι πέραν των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, σε κάθε περίπτωση η χρηματική αποζημίωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πάυσης της γεωργικής παραγωγής της Ένωσης η οποία εγγυάται την επιστημιστική ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, είναι δε απαραίτητη για την ευημερία των αγροτικών περιοχών της Ένωσης. Ως γνωστόν, η παραγωγή της Ένωσης ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και αηφόρου παραγωγής. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επιβληθούν στις εισαγωγές πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται στην Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί αφενός ότι οι αγρότες της Ένωσης θα ανταγωνίζονται επί ίσης όρης και αφετέρου ότι θα προστατεύονται αποτελεσματικά οι πολίτες, οι καταναλωτές της Ένωσης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίη η αποτελεσματικότερη έλεγχη επί των εισαγωμένων προϊόντων στα σύνορα της Ένωσης. Δυστυχώς, η Κομισιόν δεν φαίνεται πρόθυμη να απαιτήσει στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών την επιβολή ισοδύναμων προτύπων για τα, εισαγόμενα αγαθά. Σε κάθε περίπτωση στις ελόγω συμφωνίες θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον από τους εταίρους μας η συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις και προδιαγραφές και πρότυπα. Θέλω παράλληλα να υπογραμμίσω την ανάγκη προώθησης των επιθετικών συμφερόντων της Ένωσης δεδομένου του ευρέως εξαγωγικού δυναμικού, των υψηλής ποιότητας γεωργικών ειδών διατροφής της Ένωσης, το οποίο όμως υπονομεύεται από πλήθος μη δασμολογικών εμποδίων που επιβάλλουν οι εταίροι μας, οι εταίροι στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ως προς διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα, η Κομισιόν έχει προβεί σε μια εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά, σε ένα offer στο γεωργικό τομέα, ενώ το πλέον πρόσφατο κείμενο που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, αναφέρομαι στα draft modalities για τη γεωργία το 2008, θα σήμαινε σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους της ΕΕ. Η Επιτροπή η Κομισιόν καλείται να συμμορφωθεί αυστηρά με τη διαπραγματευτική εντολή που έχει λάβει από το Συμβούλιο και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην αναλαμβάνει, να μην αναλάβει εσδήποτε δεσμεύσεις που θα προκαθόριζαν τις αποφάσεις και τις αποφάσεις μας για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013. Υπογραμμίζω όλος ιδιαίτερος ότι παραχωρεί στο γεωργικό τομέα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών θα πρέπει να συνδέονται με τις ενδεχόμενες παραχωρήσεις οι οποίες θα προκύψουν από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του γύρου της Δόχα. Τέλος, η αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης από τους εμπορικούς μας εταίρους πρέπει να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες τόσο σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα στις αγροτικές διαπραγματεύσεις όσο και σε επίπεδο άκτα ως ουσιώδες μέρος της συμφωνίας. Τέλος, επισημαίνω ότι σε διμερές επίπεδο δεν είναι ικανοποιητική η προσέγγιση που ακολουθείται, σύμφωνα με την οποία ένας συνοπτικός κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης προστατεύεται μόνο από τους εμπορικούς μας εταίρους. Μόνο ένας συνοπτικός κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης προστατεύεται από τους εμπορικούς μας εταίρους. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως μια συνοπτική εισαγωγή και θα πω και εγώ, όπως και η συνάδελφος κυρία Γέγλε, ότι τροπολογίες είναι προσδεκτές και ότι σε ό,τι με αφορά θα επιδείξω πνεύμα συνθετικό, μια δημιουργική σύνθεσης, ούτω ώστε να προκύψει στο τέλος ε, ένα καλό ισορροπημένο αποτέλεσμα ε, στο κρίσιμο αυτό θέμα που αφορά τις εξωτερικές πτυχές, την εξωτερική διάσταση τη Ευρωπαϊκή ε, αγροτικής πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαστάμκο. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ήδη έχουν εγγραφεί πάρα πολλοί. Να... Έρανς Γκαρσία ο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να, να συγχαρούμε τον κύριο Παπαστάμκο, διότι αυτό το σχέδιο έκθεσης συμπεριλαμβάνει πολλές από τις ανησυχίες και τα μελήματα που έχουν οι γεωργοί, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί όσον αφορά τις συναλλαγές και ανταλλαγές για παράδειγμα, για τη θέσπιση πολυμερούς μητρώου όσον αφορά τα προϊόντα τους, ε, όσον αφορά τις ε, κυρώσεις για μη τήρηση των κανόνων, για τους κανόνες προέλευσης, ε, για το τριγωνικό εμπόριο ή τα μέτρα προώθησης που πρέπει να εισαχθούν για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Γι' αυτό συγχαίρω τον κύριο Παπαστάμκο. Επίσης λέω ότι από την Ισπανική Αντιπροσωπεία θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Διότι συμφωνούμε ότι πρέπει να απαιτήσουμε αμοιβαιότητα και πρέπει οι απαιτήσει να είναι όμοιε για να πετύχουμε μια ισορροπία στην αγορά και να αποφύγουμε πριτανεύοντα ρόλο όσον αφορά κάποιου που εισάγουν γεωργικά προϊόντα, ιδιαίτερα από τρίτε χώρε. Κυρίω πιστεύουμε ότι σε σχέση με τις σχέσεις με το Μερκοσούρ είναι μια ευκαιρία αυτή η αμοιβαιότητα να απαιτηθεί και να την εφαρμόσουμε. Επίση είναι μια δυνατότητα που πρέπει να την δούμε σε σχέση με τη συμφωνία με το Μαρόκο. Μα λείπει το στοιχείο ότι δεν γίνεται αναφορά σε σχέση με αυτή την ε, ε, συμφωνία που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχει αρνητικέ επιπτώσει για τι ε, γεωργικέ παραγωγέ τη κοινότητα. Θέλουμε επίση να γίνεται λόγο για την τομάτα και άλλα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με τη συμφωνία με το Μαρόκο, διότι είναι μια ευκαιρία πολύ πιο πριν να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να τοποθετούμε για αυτά και να τοποθετηθούμε και για το Μερκοσούρ. Επίσης σε σχέση με τις ε, μπανάνες και τα προβλήματα που υπάρχουν, εδώ στη Ισπανική Αντιπροσωπεία θα υποβάλουμε κάποια τροπολογία ώστε να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για τις ε, ε, σχέσεις με τις τρίτες χώρες και για τις μπανάνες και τη σημασία τους και για τα λουλούδια που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις παραγωγές και εισαγωγές και είναι πολύ σημαντική η πτυχή της έκθεσης για αυτό το εδάφιο, για τα άνθη. Για την παράγραφο 22 της έκθεσης θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με το σύστημα ε, τιμής εισαγωγής ε, για τα φρούτα και οποροκυπευτικά. Εδώ θα ήθελα να διαφοροποιήσουμε κάπως για την ανάγκη να τροποποιηθεί το καθεστώς ε, τιμών εισόδου για τις ντομάτες που θα προέρχονται από το Μαρόκο. Διότι το σημερινό σύστημα έχει αποδειχθεί ότι δίνει στρεβλές καταστάσεις ε, που πολλές φορές έχουν καταγγελθεί από πλευράς των παραγωγών της κοινότητας, των κοινωτικών παραγωγών και είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα δημιουργεί προβλήματα και όταν θα τροποποιηθεί αυτό το καθεστώς θα δούμε ότι ακόμα περισσότερο θα επιζημιωθεί, θα, αποβεί εις βάρος ε, των κοινοτικών παραγωγών και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Χέραντς Γκαρσία. Μόρβεϊ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ στην προσωπική μου άποψη πρέπει να... Από την άποψη των γεωργών, των τρίτων χωρών, συχνά φτωχών χωρών, είναι πραγματικά άδικο να πρέπει να εφαρμόσουν τόσο αυστηρούς ανταγωνιστικούς όρους απέναντι σε προϊόντα που επιχορηγεί και επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντα των Ευρωπαίων Γεωργών. Είναι άδικο από την μεριά τους να μην έχουν τις ίδιες δυνατότητες εξόδου στην αγορά και πρέπει να τους βοηθήσουμε για να μπορέσουν να έχουν και εκείνοι τις ίδιες ευκαιρίες. Εάν αντίθετα σε σχέση από την πλευρά των Ευρωπαίων γεωργών και ιδίως των γεωργών των παλιών σοσιαλιστικών χωρών όπως η Ουγγαρία. Αυτοί έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση και μας λένε ακριβώς το αντίθετο. Ήδη υπάρχει μια άδικη κατάσταση. Οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στους γεωργούς που δεν τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές, ε, που δεν υφίστανται τις ίδιες απαιτήσεις όπως αυτές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, όπως ισχύει στις νέες χώρες μέλη, οι επιδοτήσεις είναι χαμηλότερες αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν στα παλαιά κράτη-μέλη. Υπάρχει καταρχήν μια Υπάρχει πάντοτε μια αδικία, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει και μια τρίτη λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδεχθεί την αρχή της, ανεξαρτη... της γεωργικής ανεξαρτησίας. Κάθε χώρα ή κάθε κοινότητα και ο χωρικός κάθε χώρας, κάθε κοινότητας πρέπει να μπορεί να παράγει προϊόντα για τη δική του αγορά. Και μετά για το διεθνές εμπόριο, εκεί απλώς θα εξάγει σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν μπορούν να παράγουν τα προϊόντα αυτά. Οπότε θα εισάγονται μόνο προϊόντα που δεν μπορούν να παράξουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, που δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν, να τα παράξουν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πιο δίκαιο. Επίσης, ε, τώρα σε αφορά την ορθή μεταχείριση και την υγεία των ζώων, το ίδιο ισχύει. Επίσης και για τους περιβαλλοντικούς όρους και εκεί είναι η πιο δίκαια αντιμετώπιση. Να μην, υπάρχουν, ε, υπάρχει σημαντική μεταφορά, μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων αυτών των προϊόντων σε άλλες χώρες. Επίσης, το εμπόριο των τροφίμων των τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο χώρες και για τις εξαγωγές χώρε και για τις εισαγωγούς χώρες. Το, εμπόριο, το γεωργικό εμπόριο αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές και πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια διατροφική ανεξαρτησία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ουγγαρία, λοιπόν, θα πρέπει οι Ούγγροι καταναλωτές να καταναλώνουν τα προϊόντα των Ούγγρων γεωργών, που είναι υγιή και καλής ποιότητας. Αυτή η αρχή, πιστεύω, πρέπει να ακολουθηθεί και στις άλλες ε, χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Μισελ Νταντένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω συνάδελφο, το συνάδελφο για την σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης το πρώτο που μου φαίνεται εξαιρετικό είναι ο τόνος, ο, σταθερός και αποφασιστικός τόνος που χρησιμοποιείται σε κάθε παράγραφο, σε κάθε εδάφιο, γιατί πιστεύω ότι υπό το φως των όσων συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδείξουν πυγμή, σταθερότητα πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχει το παράδειγμα της ζάχαρης, αυτό προβάλλουμε συνήθως. Θα μπορούσαμε να δώσουμε το παράδειγμα της μπανάνας. Στη Γαλλία έχουμε υπερπόντια εδάφη όπου η μπανανοπαραγωγή πραγματικά είναι πολύ σημαντική ε, για την επιβίωση. Ε, στις αντίλες, για παράδειγμα, ο περιορισμός της μπανανοπαραγωγής θα φέρει τον πληθυσμό σε μια κατάσταση όπου μόνο το ελάχιστο εισόδημα που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα θα είναι η μόνη λύση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε ολόκληρες περιοχές για το κέρδος μερικών συμφερόντων, μερικών βιομηχανικών ε, συμφερόντων ή συμφερόντων υπηρεσιών της Υπήρου μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, και το έχω πει και άλλες φορές στην Επιτροπή αυτή, αλλά θέλω να το επαναλάβω, ότι ο, συνοριακός, ε, ο τελωνιακός έλεγχος, ο συνοριακός έλεγχος, όσο καλός κι αν είναι, ποτέ δεν θα μας προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις για τον καταναλωτή από τον έλεγχο που γίνεται σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, κάτι που μπορούμε να το κάνουμε όταν το προϊόν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι το ξέρει αυτό ο Ευρωπαίος καταναλωτής και πρέπει να συμμετέχει και αυτός στις διαπραγματεύσεις. Να έρθω τώρα σε αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υιοθετήσαμε μια τροπολογία στο άρθρο 30 του κειμένου για τις σχέσεις μας με την Νότιο Αμερική το οποίο καθορίζει την κοινή, το, το ανάτατο όριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η πρόταση του ενός συναδέλφου απορρίφθηκε. Επρόκειτο για έναν επανακαθορισμό της εντολής. Πιστεύω ότι η συζήτηση που γινόταν στα παρασκήνια του Κοινοβουλίου δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχουν απομακρυνθεί πολύ, είναι εντελώς αποσυνδεδεμένοι από την γεωργική παραγωγή. Δεν γνωρίζουν την καινούργια ισορροπία που έχει επέλθει με την είσοδο των νέων 12 κρατών μελών. Νομίζω λοιπόν ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να το ξαναθέσουμε το θέμα ε, επιτάπητος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ.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 και να υλοποιηθούν αυτοί οι όροι. Αυτό σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται σε ανταγωνισμό με παραγωγούς που δεν υλοποιούν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για την τροφική ασφάλεια. Έχουμε κοινούς κανόνες και κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει όλοι να τηρούν. Μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή και διμερός θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις και μπορούμε ίσως μέσα στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων να καθορίσουμε ποιο επίπεδο θα πρέπει να τηρείται. Όμως, τούτων λεχθέντων, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλους τομείς, άλλα πεδία όπου de facto δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες και κανονισμοί που θα μπορούσαν να ελέγχονται. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την προστασία των ζώων την ευημερία, την ευζοία των ζώων. Εκεί πρέπει να διαπιστώσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν κοινέ διατάξεις, κοινοί κανόνες και κανονισμοί για την common ε, animal welfare, δηλαδή την ευζοία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να προβληματιστούμε κάπως, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση να μας προβληματίσει αυτή η κατάσταση σε αυτό το πλαίσιο, διότι αν καθορίζουμε κάποια, κάποιες προδιαγραφές που θα, να ελέγχουμε, θα μπορούμε να ελέγχουμε στη συνέχεια, θα είναι ελέγξιμες και παληθεύσιμες, τότε θα ήταν πολύ πιο απλό να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις για το δίκαιο εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πόλσεν. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα όπως και ο Μισελ Νταντέν να πω ότι είναι πολύ καλό το κείμενο και ότι θα μπορούσα να το συνυπογράψω χωρίς κανένα πρόβλημα και με τα δύο χέρια. Ίσως βέβαια χρειάζονται ορισμένες αποσαφηνήσεις, ιδιαίτερα για τον όγκο του διεθνούς εμπορίου, γιατί γίνεται λόγος εδώ για το διεθνές εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο 8% των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνονται διεθνώς. Άρα το διεθνές εμπόριο αυτών των προϊόντων είναι πολύ μικρό τμήμα δεν μιλάω για μέσα στην Ευρώπη, μεταξύ υπήρων. Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα επί του οποίου θα μπορούσαμε ίσως να επιμείνουμε λίγο παραπάνω, ο ρόλος ορισμένων επιχειρήσεων που δεν παίζουν το παιχνίδι. Παραδείγματο χάρη επιχειρήσεις που μεταλλεύονται τις διεθνείς συνθήκες για να εγκατασταθούν εδώ ή εκεί για να κερδίσουν μερίδια αγοράς με τρόπο αρκετά δυσάρεστο, ας πούμε η Tyson που εγκαθίσταται στη Βραζιλία γιατί ξέρει ότι προβλέπεται συμφωνία με την Ευρώπη επίκειται και προλαβαίνουν, γράφουν ότι θέλουν να έχουν ένα είδος αεροπλανοφόρου εξαγωγών προς την Ευρώπη από εκεί. Το κάνουν με τα πουλερικά όπου ο τομέας απειλείται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα λέμε. Έχετε δίκιο που επιμένετε για τη ζάχαρη, όπου υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και όπου η Διεθνή Συμφωνία, η Συμφωνία με την Νότια Αμερική δείχνει ότι το Περού εποφελείται από μια ποσόστοση εξαγωγής και δεν παράγει πλέον ούτε ένα κιλό ζάχαρη. Ποιον ωφελούν λοιπόν όλα αυτά. Τέλος, σας συγχαίρω επίσης για το θέμα της μπανάνας, γιατί και αυτό το θέμα και των Καναρίων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει πια να σταματήσουμε την παλαιά λογική που ξέρουμε ότι δεν, αποφέλει, δεν ωφελεί τους γεωργούς της Γουατεμάλας και άλλων τέτοιων χωρών, αλλά μόνο τους μεγάλους παραγωγούς. Τέλος, σωστά λέτε για τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών, τις εμπορικές σχέσεις, αλλά το έλλειμμα οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή πρωτεϊνών, φυτοπρωτεϊνών για ζωοτροφές και το θέμα είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους. Θα μπορούσαμε να πούμε δυο λόγια εκεί μέσα στα πλαίσια των εμπορικών. Τα άλλα θα τα θέσει ίσως ο κύριος Άουσλινγκ στην εκθεσή του. Αλλά το θέμα του ισοζυγίου είναι κάτι το σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιωζέ. Ο Τζέιμς Νίκολσον έχει το <coughs> λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παπαστάμκο για μια πάρα πολύ έκθεση. Νομίζω έρχεται στη σωστή χρονική συγκυρία, όπου μπορούμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα από την κοινοβουλευτική μας Επίτροπη σε όλους όσους ακούν και αφουγκράζονται. Όπου και να πάει κανείς ε, στις ε, ΗΠΑ, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπου και να ταξιδέψει κανείς, όλοι θέλουν να μπουν στις αγορές μας. Γιατί, διότι <clears throat> είναι μία από τις καλύτερες και πιο κερδοφόρες παγκόσμια. Έχουμε μία κατάσταση και αναφέρεται σε αυτήν ο εισηγητή όσον αφορά την ανάπτυξη και το μέλλον και οτιδήποτε συμβεί στι διαπραγματεύσει με το Μερκοσούρ ως προς αυτά και όποιο δει αυτά τα θέματα και ξέρει κάτι για αυτά, γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει την ε, αγροτική βιομηχανία στην Ευρώπη. Δεν έχουν το ίδιο κόστος εκεί, δεν έχουν τον ίδιο ανταγωνισμό. Σίγουρα δεν έχουν ε, πολύμορφη συμμόρφωση την οποία πρέπει να, με την οποία πρέπει να ευθυγραμμίζονται όπως εμείς και απλά και μόνο αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εκεί ως όροι και προϋποθέσεις. Δεν είναι συγκρίσιμα λοιπόν τα στοιχεία αυτά μεταξύ μας. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Και αν και πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να το πούμε σαφώς αυτό ότι κάποιες, νομοθεσ... κάποιες νομοθετικές διατάξεις και οδηγίες που υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφωνόμαστε με αυτές, αν δεν υπάρξει κάτι αντίστοιχο τότε δεν μπορούμε να ε, αναμένουμε κάτι το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις διατάξεις ε, και θα εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το, το τελικό συμπέρασμα. Υπάρχει ο ΠΟΕ και θα έχουμε σίγουρα ε, το θέμα αυτό το οποίο θα τεθεί και επανειλημμένα διότι στο τέλος τέλος πρέπει κάτι να γίνει σε σχέση με αυτό το τελικό συμπέρασμα. Ε, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε από την άλλη πλευρά ότι εκείνοι από εμάς σε σχέση με την Ευρώπη που εκπροσωπούν τις ε, βιομηχανίες και τους βιομηχανικούς κύκλους και πραγματικά εδώ θέλω να αμφισβητήσω την ηθική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιείται μια άδεια του 1999 για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με τη Μερκοσούρ και μετά να έχουν το θράσος να έρχονται στην, Ευρωπαϊκή, στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να πούν υπάρχει άδεια να γίνει αυτό. Κάτι το οποίο έγινε το 1999 με 15 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν υπήρχε ακόμα το ευρώ και πάρα πολλά έχουν αλλάξει μεταξύ με 27 κράτη-μέλη. Ε, τότε πρέπει να πω ζητώ συγγνώμη λυπούμε αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει με αυτή την άδεια του 1999 και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα που τοποθετήθηκε σχετικά με αυτό, διότι ψηφίσαμε και εγώ υπεψήφισα αυτή την πρόταση. Όμως ε, η πλειοψηφία των μελών αυτού του Ευρωκοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο δεν είχαν ιδέα για την τροπολογία την οποία ψήφιζαν. Γιατί αν το γνώριζαν δεν θα ψήφιζαν όπως ψήφισαν, θα ψήφιζαν διαφορετικά. Τώρα, μακροπρόθεσμα μπορεί αυτό να επανορθωθεί βέβαια, διότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Όμως ε, σε σχέση με τη στάση που υιοθετείται σε σχέση με όσους εκπροσωπούν την ε, βιομηχανία ε, των γεωργικών προϊόντων. Το να πει κανείς ότι κάτι είναι πιο σημαντικό από τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, πιο σημαντικά από την, ε, τα γεωργικά προϊόντα. Λυπούμε, δεν είναι πιο σημαντικά αυτά από το να παράγει κανείς όπως πρέπει τα γεωργικά προϊόντα. Και πρέπει εκπροσωπώντας την γεωργία να θέσουμε τα θέματα αυτά στη σωστή τους θέση και να μην δεχτούμε να ανατρέπονται. Και επίση πρέπει να πω ότι ε, έχει επέθει ο κόρος πλέον σε σχέση με το να κατηγορούνται όλοι οι ανταγωνιστές όταν κάτι πάει στραβά. Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι οι ίδιοι πολύ πιο ενεργοί και να ε, υπερασπίζονται την ε, ε, γεωργία. Δεν είναι μόνο οι πηχαίοι τίτλοι στις εφημερίδες, κάτι πρέπει να γίνει ώστε να μπορεί να εκπροσωπείται ο κύκλος αυτός. Θα είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και αν εμείς δεν υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές διαδικασίες κανείς δεν θα το κάνει, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Ο George Λάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίσης και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παπαστάμκο για την έκθεσή του. Δεν είμαι 100% βέβαιος. Σε ποιον αναφερόταν ο συνάδελφος κύριος Νίκολσον πιο πριν για κάποιους εκπροσώπους. Ήταν όμως ε, μια, ένα παθιασμένο επιχείρημα αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα αυτής της έκθεσης, ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις με την Μερκοσούρ. Σε αυτή την έκθεση θα έλεγα υπογραμμίζονται το ότι αυτά τα οποία έχει υιοθετήσει ή έχουν διακριβωθεί για τις διαπραγματεύσεις ε, με τη Μερκοσούρ βρέθηκαν από τον τύπο, από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξε κάποια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εμπλακεί το Κοινοβούλιο και αυτό κρίμα είναι γιατί στο μέλλον θα πρέπει πραγματικά να γίνονται τα πράγματα διαφορετικά Πρωτού ανακαλύψουμε πάλι από τα μέσα ενημέρωσης ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο πάλι. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω ότι η συμφωνία Mercosur που όπως εγώ τα βλέπω τα πράγματα θα βασίζεται σε 400.000 τόνους βόηου κρέατος που θα εισάγεται στην Ένωση. Αν όλα αυτά ισχύσουν, ιδιαίτερα για τους ε, παραγωγούς, βοήου κρέατος στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στη Σκοτία, θα είναι ε, σοβαρό πλήγμα. Και η ανησυχία μου είναι ότι σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ επικεντρωνόμενοι σε κάποια θέματα μπορεί ίσως να αγνοήσουμε αυτό και στο τέλος δεν θα έχει ε, νόημα να γίνει κάτι ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ένα ε, αηφόρο μέλλον για αυτή την παραγωγή στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν η έκθεση αυτή να πάει λίγο πιο πέρα από αυτό το πλαίσιο, να ζητήσει να υπάρξει ένα impact assessment, μια μελέτη επιπτώσεων και νομίζω ότι στο 25 πρέπει να ενδυναμώσουμε. Πρέπει να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων που θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δυνατόν νωρίτερα και να υποβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο να δούμε ήδη μαύρο-άσπρο ποιε θα επιπτώσεις θα υπάρξουν από κάποια τέτοια μέτρα. Γιατί νομίζω εδώ σε σχέση με τα όσα έχουν ε, συζητηθεί και όσα πρόκειται να ε, ρυθμίσουν αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Είναι απόλυτα σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ε, να σταθμίσουμε και να κρίνουμε τι θα γίνει και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα σε σχέση με την εντολή των που δίνεται στους ε, διαπραγματευτές αν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ή όχι. Το δεύτερο αίτημά μου θα ήταν για μια μεγαλύτερη σαφήνεια να δούμε σε ποιο βαθμό και κατά πόσον μπορούν να έχουν περιθώριο για αυτές τις διαπραγματεύσεις οι διαπραγματευτές με τρίτες χώρες. Τι μπορεί να, ε, πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν και τι μπορεί να γίνει και ποια προστατευτικά μέτρα μπορούν να υιοθετηθούν για να πετύχουμε να ε, δούμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θα ισχύει ε, για την Ευρώπη. Και νομίζω θα πρέπει λοιπόν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλιστεί ότι θα ενημερωνόμαστε στο μέλλον και όχι θα να ανακαλύπτουμε από τον τύπο τέτοια στοιχεία. Να γίνει λοιπόν μια μελέτη επιπτώσεων των δυνατών ταχύτερα ώστε να ξέρουμε τι θα γίνει στην ευρωπαϊκή αγορά για την ευρωπαϊκή γεωργία και να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, αποσαφήνιση του περιθώριου για τις διαπραγματεύσεις που οι διαπραγματευτές ε, θα ε, διεξαγάγουν ε, όσον αφορά τα θέματα από την Ευρω... για την παρουσίασή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω και μπορεί αυτό και με κάποιες ε, τροπολογίες να κατατεθούν στην Επιτροπή μας για να διασφαλιστούν αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, George. Ο κύριος Ντές έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ θερμά και τον Γεώργιο Παπαστάμκο για το ότι ανέλαβε αυτό το σημαντικό θέμα και το εξεπώνησε με την έκθεσή του. Ξέρω ότι έχουμε έναν ικανότατο μαχητή για τα συμφέροντά μας στην Επιτροπή Γεωργίας με τον κύριο Παπαστάμκο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου την προηγούμενη εβδομάδα την τροπολογία την υπερψήφισαν που είχε κατατεθεί από 77 ευρωβουλευτές. Πολύ συνειδητά ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία για να μπορούμε να δούμε ποιος υπερψήφισε αυτό το αίτημα μαζί μας για πρώτη φορά ζητήθηκε αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να απαιτείται ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των ζώων και τις κοινωνικές ελάχιστες προδιαγραφές θα τηρούνται. Δεν γνωρίζω μια τέτοια απόφαση με τέτοια πλειοψηφία και με αυτούς τους όρους να έχει υιοθετηθεί ήταν 535 συνάδελφοι ευρωβουλευτές ε, που ήταν ε, ε, παρόντες στην ψηφοφορία και εξεφράστησαν. Είναι δικαίωμά μας να ζητάμε αυτά τα πράγματα. Το λέω αυτό. Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να ισχύσουν. Αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κάνουμε αυτό και έχουμε ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τα φυτικά προϊόντα, μια ολόκληρη σειρά προϊόντων αποκλείονται από τη χρήση τους, διότι οι επαΐοντες θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία που απορρέουν από τέτοιες ουσίες. Τότε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε από τον υπόλοιπο κόσμο να εισάγονται γεωργικά προϊόντα στην Ευρώπη, όπου αυτές οι ουσίες εξακολουθούν και χρησιμοποιούνται και έτσι εισάγονται με αυτές τις ουσίες τα προϊόντα στην Ευρώπη. Διότι με αυτή την λογική, εφόσον είναι επικίνδυνα για την υγεία αυτά τα προϊόντα, δεν μπορούν να εισάγονται με τη χρήση αυτών των ουσιών. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λογική που θα μπορεί να διέπει αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό πρέπει δραστικά να απαιτήσουμε αυτό να είναι σεβαστό. Και όσον αφορά το θέμα της, ε, των διαπραγματεύσεων με την Μερκοσούρ, εδώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πολύ μεγάλο τακτικής μορφής ε, σφάλμα έκανε σε σχέση με νομική βάση προηγουμένων ετών όπως επικαλούνται έδρασαν. Όμως στην εποχή της συναπόφασης είναι τεράστιο σφάλμα να μην ενημερώνεται το Κοινοβούλιο, να μην έχει ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο, ο Επίτροπος για το Διεθνές Εμπόριο να προσέλθει στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, να προσκληθεί εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας υπεύθυνα να απαντήσει τις ερωτήσεις μας και να λογοδοτήσει. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά να είναι στην Επιτροπή, στην Επιτροπή μας στο Γερμανικό Κοινοβούλιο είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα σε βάθος και είχα τότε πει στο παρελθόν ότι ακριβώς αυτά τα ίδια πράγματα ότι όταν ζητάμε ανοιχτά σύνορα όταν περνάμε, περνώντας από τα οικόπεδα αυτών των κυρίων είχαν τους υψηλότερους τείχους ε, που προστάτευαν τις ιδιοκτησίες τους. Δεν ήθελαν να ακούν καθόλου τίποτα για ανοιχτά, ε, για διαφάνεια. Τώρα ζητείτε, ζητείτε εδώ να υπάρξουν ε, να, να μην υπάρχουν σύνορα στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να έχουμε σύνορα στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι το εμπόριο πρέπει ελεύθερα να διεξάγεται. Όμως πρέπει οι κανόνες να είναι σεβαστοί και το εμπόριο να διεξάγεται με θεμητού και δίκαιους κανόνες στο παιχνίδι αυτό και επειδή από πλευράς και εισήγηση που έχω αναλάβει, δεν μπορούμε επί μήνες τώρα σε σχέση με την ε, γεωργική πολιτική να ε, μακρηγορούμε. Πρέπει να βρούμε, να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό και να υπονομεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις θέσεις. Κάτι τέτοιο θα έκανε παλιόχαρτα την έκθεσή μας και θα την καθιστούσε ανεφαξίας. Γι' αυτό πρέπει από κοινού να βρούμε μια πολύ καλή γραμμή πλεύσης και ζητούν και άλλοι συνάδελφοι να, βρούνε, να βρούμε κοινέ προδιαγραφές να ισχύουν για όλους και βρισκόμαστε στην ορθή πορεία νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άλμπερτ, συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να θυμόμαστε, το θύμισε και ο Ζόρτζ Λιόν, Lion, ότι πρέπει να έχουμε κανόνες σαφείς, διαφανείς, που να μην δημιουργούν στρεβλώσεις για να μπορέσουμε να, σε οποιαδήποτε βοήθεια δοθεί προς ε, τη Γεωργία. Ε, Γεια, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μία εκπροημίου παρατήρηση θέλω να κάνω και μία πρόταση. Εκπροημίου παρατήρηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παπασταμπό για αυτή την έκθεση. Στη σωστή χρονική συγκυρία υποβάλλεται. Έχει, έχουν συζητηθεί αυτά. Διακόπτει ο μιλητής. θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι υπήρχε λέει εντολή να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις επειδή δεν διεκόπησαν οι παλαιότερες διαπραγματεύσεις και μπορούν να συνεχιστούν τώρα μπορεί τυπικά από νομικήστική πλευρά να είναι ορθό όμως ε, δεν είναι ορθό πολιτικά εξοργίστηκα με αυτό για το ε, πόσο ελαφρά την καρδία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμφέροντά μας τα ποδοπάτησε και τα παρέκαμψε και δεν το θεώρησε αναγκαίο να μας ενημερώσει. Και γι' αυτό πρέπει πολιτικά να τοποθετηθούμε επ' αυτού και να πούμε κάθετα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούστε κύριε υπάρχει ακόμα το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή Γεωργίας που προβληματίζεται για αυτά και είναι απλό τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας να προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο και να τα λάβετε υπόψη αυτά τα στοιχεία. Τώρα, θα ήθελα να πω, εμείς πρέπει με σαφήνεια να πούμε ΠΟΕ εγώ πάντα προτιμώ διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, βρίσκονται σε εξέλιξη υπό το πλαίσιο του ΠΟΕ και ολοκληρώνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διότι, διότι όλα όσα γίνονται πολυμερός ή διμερός, διεθνώς πολυμερός ή διμερός, μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα. Ή, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες χώρες ή ομάδες χωρών σε αυτόν τον κόσμο που τα συμφέροντά τους γεωργικά πολιτικά είναι όταν θα έχουν υλοποιηθεί τότε δεν ενδιαφέρονται για τα υπόλοιπα θέματα, κλείνει το θέμα για αυτές τις χώρες. Εδώ υπάρχει κίνδυνος με αυτή την κατάσταση. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταιριάζει αυτό στην εικόνα του Μερκοσούρ. Μπορεί αυτό να ταιριάξει με το συνολικό οικοδόμημα του ΠΟΕ. Και τελευταία παρατήρηση. Πάντα οργιζόμουν, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Προς έκπληξη όλων, πρέπει να πω, από άλλους συναδέφους από το Ευρωκοινοβούλιο, επανειλημμένα θα έλεγα το παραμύθι ε, διαδίδεται στην Ευρώπη ότι με τις επιδοτήσεις που δίνουμε για τις εξαγωγές εμείς είμαστε υπεύθυνοι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Και εδώ θα ήθελα να το αποσαφηνίσω αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι επιδοτήσεις στις εξαγωγές δεν υπάρχουν πια de facto. Δεν υπάρχουν πια. Έτσι αυτό το επιχείρημα είναι αβάσιμο. Απόλυτα βάσιμο. Τελευταία παρατήρηση. Η τελευταία αυτή η παρατήρηση πρέπει να βρίσκεται υπό τον τίτλο εντιμότητα. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η γεωργική πολιτική είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινείται. Κάθε μπλοκ έχει το δικαίωμα να παράγει τέτοιον όγκο τροφίμων ώστε τους κατοίκους ε, του ή τους κατοίκους της να μπορεί να τους ε, τρέφει επαρκώς. Και κατά τα άλλα, από την, για την ανταλλαγή απόψεων, μπορούμε, α, ανταλλαγή προϊόντων και τις συναλλαγές μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε τις διαφορετικές πτυχές. Έχουμε έναν καλό εταίρο με τον ε, κύριο Παπαστάμκο και αυτά μπορούν να προωθούν. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση που κάνουμε να καταστεί σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι οικονομικές πολιτικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις πρέπει να διεξάγονται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι εν κενό. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Γιάρα. Η Ελίζα Πεθιγέγκο πρέπει να φύγει, επομένω θα της δώσουμε το λόγο τώρα. Η ε, κυρία Γέγκλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προαναφέρθηκαν, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Και τώρα, ακριβώς πιο πριν, είχα μια συζήτηση με τον Καναδό πρέσβη και την, το Σάββατο θα πάω στον Καναδά, θα πετάξω με αεροπλάνο και στον Καναδά θα με ξαναρωτήσουν και σε μεσαφήνεια θα μου πούν ότι για τη συμφωνία Καναδά Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται καθοδόν προς την ορθή κατεύθυνση. Ο πρέσβης είπε ότι βρισκόμαστε τώρα στα δύσκολα θέματα και το δύσκολο θέμα είναι η γεωργία. Πρόκειται για το κρέας, εισαγωγή κρέατος, εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και ε, ονομασία, ε, γεωγραφική ονομασία προέλευσης. Αυτά είναι τα δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσημα δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα όμως για όλα αυτά. Στο τέλος θα πρέπει να μπορέσουμε να εγκρίνουμε ως κοινοβούλιο να απορρίψουμε. Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας θα ήθελα να το απορρίψουμε, αλλά για την απόρριψη δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε πλειοψηφία στην Ολομέλεια, γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποιε λύσει και κάποιου συμβιβασμού. Γι' αυτό υποστηρίζω την έκθεση Παπαστάμκου. Και σε αυτό το σημείο πρέπει ακόμα πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια να δούμε πώ μπορούμε να απαιτήσουμε να μπορούμε σε τέτοιε διαπραγματεύσει έγκαιρα να εμπλεκόμαστε. Ποιο θα μα πει και θα μα λέει ποια είναι η εντολή διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων και πώ μπορούμε να απαιτήσουμε η Ευρωπαϊκή Γεωργία με όλε αυτέ τι συμφωνίε που θα αρχίσουν να λειτουργούν θα μπορέσει να ληφθεί υπόψη τα γαλλικά νησιά ακριβώς μπροστά από τον Καναδά. Σαν ε, Πιέρ και Μικελόν για τα θέματα αλληλείας. Μας παρακάμπτουν όμως και έχω την εντύπωση ότι δεν κάνουν τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εδώ επαρκούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο ματό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη ότι καθυστέρησα σε σχέση με την Επιτροπή Αλίας. Είχαμε, για την Αλία είχαμε ψηφοφορίες. Και πολύ σύντομα λοιπόν θα ήθελα να πω συγχαίρω τον κύριο Παπαστάμκο, είναι μια έκθεση πλήρης, μια έκθεση που πραγματικά έχει επίπτωση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Διαπραγματεύσεις που δυστυχώς για τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το γεωργικό τομέα ήταν πάντα αρνητικές. Σκέφτομαι την Κολομβία, έχω υπόψη το Περού. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και το Μερκοσούρ σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ξεκινούν κάποιες διαπραγματεύσεις και μετά στη συνέχεια υπό το γεωργικό πρίσμα της γεωργίας πρέπει να ζητούνται αποζημιώσεις ή αντισταθμίσεις ή να ζητηθούν ρήτρες ασφάλισης ή διασφάλισης διότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις λαμβάνοντας υπόψη ένα τομέα τόσο σημαντικό όπως τον τομέα της γεωργίας. Είναι θεμελιώδες λοιπόν αυτό να τονίσουμε αυτό το θέμα όπως το κάνει η έκθεση Παπαστάμκου να μην ξεκινήσουν οποιασδήποτε μορφή διαπραγματεύσει χωρί προηγούμενη αποτίμηση, εκτίμηση επιπτώσεων, μελέτη επιπτώσεων. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτά ε, με τροπολογίε πρέπει να καλύψουμε ένα θέμα το οποίο δεν καλύπτεται για τα Κανάρια νησιά και τι απομακρυσμένε περιοχέ, ε, όπω είναι η μπανάνα. Συνεχίζεται ο πόλεμος τη μπανάνας ε, και πρέπει γι' αυτό να συμπεριληφθεί το θέμα των μπανανών στην έκθεση αυτή. Είναι θεμελιώδες αυτό το στοιχείο. Και από την άλλη πλευρά και στι με το Μαρόκο πρέπει να γίνει κάποια αναφορά. Όχι επειδή είμαστε εναντίον αφεαυτού, αφεαυτής αυτής συμφωνίας με το Μαρόκο. Σε αυτή τη συμφωνία με το Μαρόκο πρέπει να γνωρίζουμε με σαφήνεια δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Αυτό δεν είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό που ε, θεσπίζει και διαμορφώνει τι τιμέ εισαγωγέ. Γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει κάποια αναφορά σε αυτή την πτυχή, σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάτο. Μάια Chairman. Ευχαριστώ κύριε Θέλω και εγώ να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή γιατί δεν είχα έρθει από την αρχή της συζήτησης γιατί συζητούσα με τις κλιματολογικές αλλαγές αλλού και ε, τις συνομιλίες του Μερκοσούρ τις ανέφερα και εγώ εκεί γιατί πράγματι αν θέλουμε μια συμφωνία που να καταστρέφει την παραγωγή βοήου κρέατος στην ε, Ένωση θα αναγκαστούμε να εισαγάγουμε περισσότερα και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την ευθεία γλώσσα του εισηγητή και την ειλικρίνειά του. Νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί από προηγούμενες ψηφοφορίες, όπως είπε και η κυρία Γέγκλε, η έκθεση Σαλαφράγκα ζητούσε, δεχόταν τις συνομιλίες του Μερκοσούρ αλλά χωρίς να αναφέρει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι διμερείς συμφωνίες στην πολιτική της Ένωσης. Ενώ αυτή η έκθεση συνδυάζει όλες μας τις ανησυχίες πολύ σωστά και το μήνυμα προς την Κομισιό νομίζω θα το έχει καταλάβει πια εκείνη γιατί είναι αλήθεια ότι έχουν περιφρονήσει το Κοινοβούλιο και οι απαντήσεις που έχουμε λάβει γραπτός αλλά και προφορικός στην Ολομέλεια ήταν ασαφέστατες όλες και μάλλον στόχευαν σε καθυστερήσεις παρά σε πραγματική απάντηση και ανταπόκριση των ανησυχιών των πολιτών μας. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την έκθεση, δεν ξέρω αν χρειάζεται και πολλές αλλαγές γιατί νομίζω ότι είναι σαφέστατη και η ιδέα μιας μελέτης αξιολόγηση αντικτύπου είναι πολύ ουσιώδης ελπίζω να στηριχθεί όπως θα έπρεπε, όχι μόνο εδώ από την Επιτροπή μας, αλλά και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μαγκίνες. Ο κύριος Ντότς έχει το λόγο. Thank you. Uh, Κυρία Ντότς, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα είχα μια σειρά συναντήσεων με γεωργούς σε όλη την Βόρειο Ιρλανδία και κάτι που τους καταθλίβει ιδιαίτερα είναι ότι στη διάρκεια όλων αυτών των διαπραγματεύσεων η γεωργία θεωρείται πάντοτε ως ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης που πρέπει πάντοτε να κάνει θυσίες εις όφελος άλλων κλάδων. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση έρχεται και το αναγνωρίζει αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα εκφράζει ένα, ένα συνέστημα που το βλέπω πολύ συχνά στην πατρίδα μου. Επίσης, να πω ότι στηρίζω έντονα το σημείο 2. Η ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων στην Ευρώπη είναι επιταγή της κοινωνίας μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα όργανα πρέπει να το διασφαλίσουν αυτό. Άλλες χώρες όπως η Κίνα αυξάνουν τη δυνατότητά τους να διασφαλίσουν τις ε, την ασφάλεια των τροφίμων για τις επόμενες γενναίες. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη. Τώρα, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Πρέπει να ε, διακρίνουμε μεταξύ την ανάγκη της προστασίας και της δικαιοσύνης για τους ε, γεωργούς μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης που ίσως να μην είναι επιταγές σε τρίτες χώρες, να μην υφίστανται σε τρίτες χρόνες. Συμφωνώ και επαναλαμβάνω τα σχόλια των συναδέλφων για τις διαπραγματεύσεις. Ο τομέας του βόηου κρέατος στη Βόρειο Ιρλανδία διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο και ίσως γίνουμε παραχωγός υψηλής ε, ποιότητας με ιχνηλασιμότητα. Ε, αυτοί οι κανόνες ε, επεκτείνονται στον τομέα του χείριου κρέατος και των πουλερικών. Νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να έρθει στην Επιτροπή μας και να μας εξηγήσει τις προθέσεις της και να κάνουμε μια διεξοδική μελέτη αντικτύπου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Λουίς Κάμπολα Σαντόσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παπαστάμκο για την δουλειά του που πραγματικά αντανακλά τις ανησυχίες μας. Θα ήθελα μόνο να σας ενημερώσω για κάτι. Ανήκω στην, αντιπροσω... στην διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με το Μέρκοσουρ και έχουμε κάνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, παρουσία του... Ε, πρέσβεως της Βραζιλίας, ο οποίος διευθύνει τον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή μια μελέτη αντικτύπου, όχι μόνο για το γεωργικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς. Για, την για, να συζητηθούν όλα τα υπέρ και τα κατά. Όλοι έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η γεωργία βρίσκεται υποπίεση. Προφανώς η Ευρώπη πραγματικά επιθυμεί το άνοιγμα των αγορών γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στην εξαγωγή και άλλων γεωργικών προϊόντων. Εμείς βρισκόμαστε εδώ ως προασπιστές της γεωργίας. Ακόμα πιο δύσκολος ο ρόλος μας γίνεται στο πλαίσιο αυτό. Σημερίζομαι τις ανησυχίες του συναδέλφου Παπαστάμκου. Ευχαριστώ, Λουίσα. Παντάου Νέβες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη από τον Πρόεδρο και από τους άλλους συναδέλφους γιατί ήρθα με μια μικρή ε, καθυστέρηση. Ήμουνα στην Επιτροπή Αλίας όπου γινόντουσαν ψηφοφορίες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να μην παρέμβω όταν συζητείτε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ο συνάδελφος Παπαστάμκος ε, ε, θα ήθελα καταρχήν να το συγχαρώ βέβαια για το περιέχον, ε, το πολύ περιεκτικό που μας παρουσίασε και εξάλλου υπήρξε και πολύ σαφής. Ε, ζητώ συγγνώμη για την φύση της παρέμβασής μου. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές εμπόριο αποτελεί ίσως ε, ε, τη χειρότερη νόμιμη απειλή για την ευρωπαϊκή γεωργία σε μια κατάσταση όπως η σημερινή, που είναι πάρα πολύ δύσκολη για τόσους κλάδους που διέρχονται μια σοβαρή κρίση και μπροστά σε ένα μέλλον το οποίο δεν φαίνεται και ιδιαίτερα ρόδινο, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τον προϋπολογισμό για την ΚΑΠ μετά το 2013, έχω πραγματικά την εντύπωση ότι Παρόλο που οι γεωργοί μας κάνουν ό,τι μπορούν, ε, επενδύουν, ε, κάνουν αμοιβέ συμφωνίες, ε, βρουν τρόπους εγγύησης της αηφόρου ανάπτυξης, πρέπει να υποστούν τις συνθήκες της κάθε συμφωνίας με το Μέρκοσουρ, με το Μαρόκο ή δεν ξέρω εγώ με ποια άλλη χώρα μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρξε κάποια σωστή, προσεγμένη, ε, κάποιος συγκεκριμένος προσεγμένος προγραμματισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητούμε από τους γεωργούς μας ταυτόχρονα να προσαρμόζονται στις ε, σημερινές και στις μελλοντικές συνθήκες της γεωργίας και από την άλλη ταυτόχρονα και ξαφνικά να τους τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια δημιουργώντας νέους κανόνες παιχνιδιού με τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστούν. Είναι πάντοτε μια δυσμενής θέση στην οποία περιέρχονται, γιατί οι ζημίες, οι επιπτώσεις για τους γεωργούς μας είναι πιο σοβαρές ακόμη. Σε, σε σχέση με όλους τους άλλους οι οποίοι εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Αρμόδιο Επιτροπό για τη Γεωργία ε, τα θέματα του ανταγωνισμού δεν, δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά τα θέματα ανταγωνισμού έχουν ε, σοβαρότατες συνέπειες για τη γεωργία. Και είναι ένας άνισος αγώνας αυτός ε, που οι γεωργοί μας πρέπει να διεξάγουν και να νικήσουν κιόλας. Στο πλαίσιο αυτό, καλό θα είναι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ότι ό,τι κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει σημαντικότατο αντίκτυπο. Μιλούμε για το άδειασμα των ε, περιοχών της υπαίθρου από τον πληθυσμό τους, για κοινωνικές συνθήκες που χειροτερεύουν, ε, για τις δυσκολίες του εφοδιασμού, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα ακούμε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Η γεωργία λοιπόν δεν είναι μόνο καθαρά γεωργία, αλλά έχει προεκτάσεις και σε πολλούς άλλους τομείς. Ίσως ε, λέω πράγματα που έχουν πει και άλλοι, αλλά θα ήθελα να τονίσω τρεις πτυχές που τις θεωρώ ζωτικής σημασίας και οι οποίες ε, ήδη εμφανίζονται στην έκθεση. Καταρχήν, όλα τα προϊόντα τα οποία θα φτάσουν, θα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρούν με ακρίβεια και αυστηρότητα τις ίδιες, τους ίδιους κανόνες παραγωγής που επιβάλλουμε στους γεωργούς μας. Δεύτερον, η αξιολόγηση των αντιπτώσεων. Το είπε ήδη ο συνάδελφος Κάπολος Άντος. Ναι, γίνεται αυτή η μελέτη ε, αντικτύπου επιπτώσεων, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ε, σε μια συνάντηση των βουλευτών ε, των ε, με, α, α, πολύ απομακρυσμένων περιοχών, ο πρόεδρος Μπαρόσο ζήτησε να μην γίνουν ποτέ δεκτές συμφωνίες ε, στη Γεωργία χωρίς να γίνεται αξιολόγηση επιπτώσεων. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε ότι πάντοτε θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει περισσότερο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε πάντα να παραμεριζόμαστε. Δεν μπορούμε πάντοτε να υφιστάμεθα τις συνθήκες χωρίς να έχουμε μπορέσει να συμβάλλουμε με χρήσιμο τρόπο. Πρόεδρος, κλείνω αυτή τη σειρά παρεμβάσεων. Ο κύριος Τζοβάνι θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο Παπαστάμκο για την πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία μάλλον θα πρέπει και αυτά να ενταχθούν στην έκθεση. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, παράλληλα με την εργασία που γίνεται εδώ, συζητούν, συζητώνται αντισταθμιστικά μέτρα για τις μπανάνες. <laughs> Θέμα που ανέφερε εν συντομία και ο συνάδελφος Μάτο. Και είναι φανερό ότι τα τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα ε, στην κατάσταση την τρέχουσα τις διαδικασίες προϋπολογισμού δεν θα μπορέσουν να προβλεφθούν για το μέλλον. Ε, σε αυτή την αναθεώρηση προς τα κάτω του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά κράτη-μέλη και το Συμβούλιο σήμερα μας ζητούν να προβλέψουμε καινούργιες συμφωνίες που μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τη γεωργία δεν μπορούμε σε αυτές τις καινούργιες ε, συμφωνίες να έχουμε αντισταθμιστικά μέτρα, ε, μέτρα αποζημιώσεων, ε, είτε με το Μερκοσούρ είτε με το Μαρόκο. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι λοιπόν κίνδυνοι για την γεωργία. Ο συνάδελφος Ντέσα πολύ καλά έκανε που μίλησε για, έκανε λόγο για μια τροπολογία που επιβάλλει την αμοιβαιότητα στις συνθήκες παραγωγής. Αλλά θέλω να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση και μεγάλη εξωτερική αξία στις, ε, στον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι συμφωνίες στη Γεωργία. Και ιδίως τι θα συμβεί στη Μεσογειακή Γεωργία ε, ε, μέσα από τη συμφωνία που προβλέπεται με το Μαρόκο. Όλος ο νότος της Ευρώπης πραγματικά θα υποστεί σημαντικότερες, πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα όσπρια στα... και στα οποροκυπευτικά. Ε, ζητώ λοιπόν εντονότατα να παρουσιαστούν δημόσια ε, τα στοιχεία από τις μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων έτσι ώστε όλοι οι βουλευτές τη στιγμή που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία όχι μόνο εκείνοι που είναι μέλη της Επιτροπής ε, Γεωργίας και πιστεύω ότι ασφαλώς θα έχουν αρνητική άποψη γι' αυτά. Αλλά και όλοι οι άλλοι βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, και στις άλλες επιτροπές να μπορέσουν με, με τα λόγου γνώσεως να ε, με, τα λόγου γνώσεως ε, να εκφράσουν ε, την συμφωνία ή τη διαφωνία τους για τις συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πολύ καλά. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Διευθυντή Σιβένας, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Γιώργο Παπαστάμκο και να προσπαθήσω να κλείσω με δύο έννοιες. Πρώτον, πιστεύω ότι η Επιτροπή μας έχει σαφέστατες και ξεκάθαρες ιδέες. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ούτε πολιτικές αποχρώσεις ούτε ερμηνείες. Θέλουμε η Γεωργία να μετράει ο λόγος της σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να μην είναι πάντοτε υποδέστερη απέναντι στους άλλους τομείς. Προφανώς δεν αρκεί η Επιτροπή Γεωργίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είμαστε αρκετοί. Πρέπει να καταφέρουμε να επιτελέσουμε ένα πολιτικό έργο και εδώ συμμερίζομαι την εξαιρετική δουλειά του Χέλμαντες στην προηγούμενη Ολομέλεια. Πρέπει να κάνουμε ένα πολιτικό έργο λοιπόν για να παρατείνουμε, να επεκτείνουμε τη συνένεση που υπάρχει εδώ και στους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ολομέλεια. Όπως, είπε, όπως λέει η έκθεση του κύριου Παπαστάμκου με πολύ σαφή τρόπο, ε, οι κανόνες, ε, καλύτεροι είναι οι κανόνες οι σαφείς, οι ξεκάθαροι που δεν δημιουργούν στρεβλώσεις παρά η οποιαδήποτε συμφωνία που θα έχουμε για την γεωργία. Είμαστε η περιοχή ε, που εισαγάγει περισσότερα προϊόντα από κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη. Προφανώς πρέπει οι γεωργοί μας να μην συνθλιβούν από τους κανόνες που εμείς βέβαια έχουμε επεξεργαστεί και έχουμε εκδώσει για τους οποίους κανόνες είμαστε φυσικά περήφανοι αλλά ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και άλλοι που εξάγουν στην Ευρώπη θα ε, τους σεβαστούν και θα τους στήρουν τους κανόνες αυτές. Υπάρχει το πολιτικό θέμα και το τεχνικό θέμα. Δίνω λοιπόν τώρα τον λόγο λόγο στον Διευθυντή Yeah. Uh, Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και τον εισηγητή για την συνοπτικότατη αυτή έκθεση, την πολύ περιληπτική. Θα ήθελα να σας πω ότι θα βασιστώ κυρίως στα βασικά θέματα που έθιξε ο εισηγητής θα μπορούσα βέβαια τις περαιτέρω λεπτομέρειες να τις κάνω άλλη φορά ή γραπτός για να σας διευκολύνω ή δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε εσείς οι ίδιοι καταρχάς. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για την Επιτροπή σας να ερχόμαστε, να σας παρουσιάζουμε, να συζητούμε όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουμε με τρίτες χώρες. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε, ποτέ. Είμαστε διαθέσιμοι λοιπόν για τέτοιου είδους ανταλλαγές. Αρχίζω από το εξή. Μιλήσαμε για τα 7 δισεκατομμύρια το έλλειμμα το 2008. Σωστό είναι αυτό αλλά το 2008 ήταν, δεν ήταν καθόλου χαρακτηριστικό έτος λόγω των τεκτενωμένων στις διεθνείς αγορές. Αν θέλουμε λοιπόν να το εξυγχρονίσουμε αυτά τα στοιχεία με τα τελευταία που έχουμε του 9, το έλλειμμα ήταν μεταξύ 2,5 και 3 δισεκατομμύρια, στο ίδιο επίπεδο δηλαδή όπως το 7. Γενικά θα έλεγα ότι τη δεκαετία του 80 όταν είχαμε τα τεράστια περισσεύματα, πλεονάσματα, το εμπορικό μας έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι εκείνο που είχαμε στη δεκαετία ε, κατά τα χρόνια από το 2000 μέχρι το 2006. Δεύτερη παρατήρηση. Σωστά τονίσατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους δασμούς για τις εισαγωγέ βοήου κρέατος αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα, δεν είναι μονομερή. Εμείς μειώσαμε τα κυρωτικά αυτά μέτρα μετά τα αντίστοιχα μέτρα των Αμερικανών. Στη Γεωργία υπήρξε μια συμφωνία που εφαρμόζουμε πάντα με τις τρίτες χώρες. Προσπαθούμε δηλαδή πάντοτε να πετύχουμε ως το δυνατόν περισσότερα για να αυξήσουμε την παρουσία ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε τρίτες αγορές. Ως παράδειγμα φέρνω την Κορέα όπου προσπαθήσαμε να μεγιστοποιήσουμε τις εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων και για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε ένα ειδικό κεφάλαιο με γεωγραφικά δεδομένα για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως ξέρετε η κορεατική αγορά είναι πολύ καλή για υψηλού επίπεδου και κερδοφόρα προϊόντα. Για τις ε, μελέτες αντικτύπου για το Μερκοσούρ το 2009 θα ενημερωθεί θα ενημερωθούν αυτά τα στοιχεία στις αρχές του 2011 και τότε θα έχετε τη δυνατότητα κι εσείς να τα εξετάσετε όσο θέλετε. Τώρα για τη ζάχαρη, δικαίως είπατε ότι είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν και προσπαθούμε όποτε χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να, να μην χρειάζεται να αλλάζουμε ή να μειώνουμε τους ρυθμούς εισαγωγών εκτός ποσοστώσεων. Θέλω όμως να πω κάτι πιο συγκεκριμένο για τα πρότυπα που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσαμε να τα επιβάλλουμε και σε τρίτες χώρες. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τα γεωργικά προϊόντα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι υποχρεωμένα να σέβονται τα πρότυπα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτά αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και προϊόντα που αφορούν την υγεία ζώων και φυτών. Διασφαλίζουμε λοιπόν ότι οι εισαγωγές αυτές συμφωνούν με τα πρότυπά μας υγείας και ασφαλείας, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις δικές μας μεθόδους παραγωγής σε τρίτες χώρες όπως την ευημερία των ζώων ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε υψηλού επίπεδου πρότυπα και είναι δικαίωμά μας αυτό, δυστυχώς δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στις τρίτες χώρες. Μπορούμε όμως τις απαιτήσει αυτές ή τα κριτήρια αυτά, τα πρότυπα, να τα ζητούμε από τους παραγωγούς μας αυξάνοντας την ποιότητα των προϊόντων μας και γνωστοποιώντας το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται σε πολύ ψηλά πρότυπα και υψηλότερα από των εισαγωμένων. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα από τους γεωργούς μας για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά Όσο για την προώθηση των συμφερόντων της Ένωσης. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω, να σας διαβεβαιώσω ότι είναι προτεραιότητά μας, όπως είπαμε σε προηγούμενη συνάντηση πριν τις διακοπές, ότι δύο τρίτα των εξαγωγών μας είναι προϊόντα μεταποιημένα υψηλής ποιότητας και αξίας. Είμαστε ίσως οι ισχυρότεροι στη διεθνή αγορά για τέτοιου είδους προϊόντα μεταποιημένα και υψηλής αξίας και ποιότητας. Θα οθήσουμε λοιπόν όσο γίνεται σε πολυμερές επίπεδο και σε διμερές επίπεδο τα προϊόντα μας. Για την προώθηση πάλι θα ήθελα να σας πω ότι εσωτερικά αυτή τη στιγμή θέλουμε να βρούμε, ψάχνουμε πώς θα βελούσαμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των δικασιών εσωτερικά και εξωτερικά. Για την Τόχα θα ήθελα να σας πω ότι αποσαφηνίσαμε παντού ότι τίποτα δεν θα γίνει δεκτό αν δεν γίνουν δεκτά όλα μαζί. Για μας αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία που να μην ανταποκρίνεται, να μην την χάνει ανταπόκριση για τις υπηρεσίες και άλλους τομείς και από τους εταίρους μας. Και θα ήθελα να σας πω ότι για μας είναι αδιανόητο να υπάρξει συμφωνία χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα ως προς τα γεωγραφικά στοιχεία και στα μητρώα και στην προστασία των τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων ανάλογη με εκείνη που εφαρμόζουμε για τα ινοπνευματώδη. Επίσης θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα γεωγραφικά στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται στο άκτα όπως είπε και ένα μέλος της Επιτροπής σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουν να υπάρχουν γεωγραφικά στοιχεία στο άκτα. Για τον κλειστό κατάλογο τώρα των γεωγραφικών στοιχείων. Όπως ξέρατε έγιναν πολλές και μακρές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη επ' αυτού και τον κατάλογο αυτών των γεωγραφικών στοιχείων τον κάναμε με τη βοήθεια, τον καταρτήσαμε με τη βοήθεια των χωρών μελών με βάση μια απλή αρχή ζητήσαμε από τα κράτη να μας πούν ποια είναι τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει όντως πραγματική εμπορική ροή με διάφορες τρίτες χώρες. Και έκαναν τις προτάσεις των και εμείς καταρτήσαμε τον κατάλογο. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι κλειστός ο κατάλογος. Οι μικτές επιτροπές μπορούν να προσθέσουν και άλλα ονόματα. Και βέβαια, αν υπάρξουν νέα προϊόντα στις αγορές των τρίτων χωρών, με μεγάλη χαρά θα τα συμπεριλάβουμε στον κατάλογο. Επίσης ακούστηκαν πολλά για το Μερκοσούρ. Δεν είμαι ειδικό για αυτή τη διαπραγμάτευση, αλλά ακούστηκε και κάτι για το Περού και τη ζάχαρη του. Uh, Α, την Κεντρική Αμερική είναι. Μα είπαν ότι το Περού δεν έχει μεγάλη παραγωγή ζάχαρη στο 2008, 900, τόνοι μόνο. Η κατανάλωση είναι ψηλότερη από την παραγωγή του, αλλά ζήτησαν στις διαπραγματεύσεις να υποθεί κάτι και για τη ζάχαρη, 32.000 τόνους και το δεχτήκαμε για να συμπεριληφθεί και αυτό στα γεωγραφικά στοιχεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί σας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση έχουμε με τρίτες χώρες ή ε, πολυμερείς διαπραγματεύσεις και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και απορίες σας και μπορούμε να σας δώσουμε και περαιτέρω λεπτομέρειες αν τις ζητήσετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας ευχαριστήσουμε τον δόκτωρ ε, Σιβένας ε, και τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας έκανε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, δεν ξέρω αν, ικανοποιήθηκαν, αν έμειναν ικανοποιημένοι όλοι οι βουλευτές από την παρέμβαση του κυρίου Σιβένας, αλλά πάντως τον ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, ανταποδίδοντας τα καλά λόγια που είπατε για την ε, έκθεση την οποία εκπώνησα, θέλω να σας πω ότι ε, αποτέλεσε πηγή έμπνευση για μένα η ανάγνωση του βιβλίου το οποίο είχατε δημοσιεύσει ε, προ λίγο καιρού και πάνω στο γεωργικό θέμα και θέλω να σας πω ότι το διάβασα με τα μεγίστης προσοχής. Ε, πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος ε, έχει περάσει, έχει παρέλθει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά τι παρατηρήσει. Θέλω να ευχαριστήσω τις συναδέλφου και του συναδέλφου για τι δημιουργικέ του συνεισφορέ, πράγματι, οι οποίε θα ληφθούν υπόψη και πιστεύω ότι θα κατατεθούν και ε, τροπολογίες από του συναδέλφου, πάντα βεβαίω, μέσα σε ένα ε, όριο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τροπολογιών. Και θα υπάρξει και πνεύμα ε, συνεννόησης και συνένεση. Ε, στην κυρία Χέραντς Γκαρσία ε, αναφέρθηκε στο τριγωνικό εμπόριο, ε, στην αμοιβαιότητα με Μερκοσούρ αλλά και με Μαρόκο. Και θέλω να πω ότι πράγματι συμφωνώ μαζί της ότι η συμφωνία με το Μαρόκο θα πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαιότητα. Αναφέρθηκε στη συμφωνία για τις μπανάνες ε, και εδώ απαντώ και στον κύριο Μάτο αλλά και στον κύριο Νταντέν. Άφησα επί χώρο για να υπάρχει ισπανική παρέμβαση στο θέμα της μπανάνας όπως εσείς ε, τη βλέπετε ορθολογικά. Ε, θέλω να είμαι απολύτως ε, ειλικρινής ε, μαζί σας, ε, γιατί ξέρω ότι το θέμα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και θέλω να το πω πολύ ανοιχτά ότι περιμένω τη δική σας συνεισφορά επί του θέματος αυτού. για την παράγραφο 22 σε ό,τι αφορά την ντομάτα, ναι, συμφωνώ και άλλωστε έχει έχουμε καταθέσει, κάνει και ερώτηση για τις ντομάτες από το Μαρόκο. Πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε, αλλά γιατί ο χρόνος πιέζει. Η κυρία Μορβάη αναφέρθηκε στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολύ σωστό. Θέλω να πω πολύ απλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ανοιχτή αγορά στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις αγωγές προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το ότι δεν ανοίγουν τα σύνορα οι ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των αναπτυσσομένων χωρών δεν βλάπτει μόνο τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστικών χωρών, αλλά βλάπτει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, το ότι οι, αντα... οι εταίροι μας ε, δεν έχουν ανοίξει την αγορά τους όσο θα έπρεπε ε, και αυτοί. Επίσης αναφερθήκατε στη διάκριση μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών, αλλά θέλω να πω ότι ε, δεν είναι αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Αυτό αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής, πολύ σωστά στην ευζοία και στο περιβάλλον και έθιξε η κυρία Μορβάη και ένα θέμα καταναλωτικού εθνοκεντρισμού, θα μπορούσα να το πω έτσι. Δηλαδή οι Ούγγροι να αγοράζουν αγγλικά προϊόντα. Ε, δεν θέλω αυτό να το σχολιάσω περισσότερο. Και ο κύριος Νταντέν αναφέρθηκε στα υπερπόντια εδάφη και στη ζάχαρη ε, και στις μπανάνες, αλλά και έκανε μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση ότι ο τελωνιακός ή συνοριακός έλεγχος δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικός ε, έλεγχος όσο είναι αυτό σε όλο το μήκος της διατροφικής ε, αλυσίδας. Και πολύ καλά έκανε αυτό που το οποίο είπε και ο κύριος Ντες που αναφέρθηκε στην παράγραφο που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για την διαπραγματευτική εντολή για το mandate. Και η κυρία Πόλσεν ε, συγκράτησα με ξεχωριστό ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις για τους κοινού κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους, για την ευ ευζοία των ζώων, αυτό που ε, για το animal welfare και την έκκληση την οποία απευθύνεται... και συμφωνώ απολύτως ε, μαζί σας. Ο κύριος Μποβέ πολύ σωστά προσδιορίσε τον όγκο των αγροτικών εμπορικών ροών στο 8% του συνολικού ε, εμπορίου και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του με την παρατήρηση της ευκαιριακής εγκατάστασης πολυεθνικών εταιριών δίκην αεροπλανοφόρων εκεί όπου ανοίγουν αγορές σε σχέση ε, δηλαδή τρίτων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστά είπατε ότι είναι εύγλωτη η περίπτωση του Περού ε, για το Ζάχαρης. Αυτό απάντησε και ο κύριος Σιβένας. Και θέλω να πω ότι, και να πω ανοιχτά τη θέση μου, κοιτάξτε, με την αναθεώρηση του το Ζάχαρης, αυτό θέλω να το ακούσει η Κομισιόν, δεν μεταφέρθηκε εισόδημα από τους Ευρωπαίους παραγωγούς υπέρ των παραγωγών των αναπτυσσομένων χωρών. Μεταφέρθηκε εισόδημα από τους Ευρωπαίους παραγωγούς υπέρ λιγοστών πολιεθνικών εταιριών. Αυτό είναι το τραγικό το οποίο έχει γίνει με την αθεώρηση του καθεστώτος ζάχαρης. Εάν η Κομισιόν φέρει στοιχεία ότι αυξήθηκε το εισόδημα φτωχών ανθρώπων τρίτων χωρών, ναι, να πούμε μεταφέρθηκε εισόδημα από εδώ υπέρ φτωχών παραγωγών σε τρίτες χώρες. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια και αυτό είναι τραγικό το οποίο συμβαίνει. Ο κύριος Νίκολσον ε, διατύπωσε την ε, επιθυμία όλων των τρίτων χωρών για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πάρα πολύ ελκυστική αγορά ε, και αυτό είναι σημαντικό και έθιξε το θέμα των προδιαγραφών, των standards και για την, ε, ξεχωριστή εντύπωση μου άρεσε η διατύπωση περιηθικής νομιμοποίησεως της Κομισιόν σχετικά με το mandate, με το μαντά, με την εντολή για τις διαπραγματεύσεις ε, με την Mercosur ε, και όπως επίσης και αυτά αφέρθηκε και ο ίδιος στην τροπολογία στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Λάιον συγκράτησα τις παρατηρήσεις του για την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Mercosur. στην εισαγωγή βοήου κρέατος, το έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι αυτό, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και συμφωνώ απόλυτα μαζί του με την ανάγκη ενδυνάμωσης παραγράφου 25, του σημείου 25 ε, της έκθεσής μου, δηλαδή ε, ζητούμε από την Κομισιό να προβεί άμεσα ε, σε, μελέτη, ε, στην αξιολόγηση του αντικτύπου, σε μελέτη των επιπτώσεων. Ο κύριος Ντέσ αναφέρθηκε και αυτό στην προφορική τροπολογία στην Ολομέλεια και στη χρήση ουσιών, αναφέρθηκε σε, σε ζητήματα φυτογειονομικού ελέγχου κατά τις αγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ίδιος επίσης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στις διαπραγματεύσει με τι χώρες Μερκοσούρ, στο ρόλο της Κομισιόν, στη στάση της Κομισιόν και στην εντολή τη διαπραγματευτική. Όπως και ο κύριο Γιάρ αναφέρθηκε στην διαπραγματευτική εντολή ε, και στα θεσμικά τρίκ τα οποία επικαλείται η, η Κομισιόν, τα θεσμικά τρίκ, συγγνώμη, ε, στις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ότι είναι και τις επιδοτήσεις μας στις εξαγωγές πράγματι δεν είναι, πολύ σωστά το διευκρίνησε, δηλαδή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στις εξαγωγές που δεν υπάρχουν, άλλες χώρες τρίτες ανταγωνιστικές χρησιμοποιούν εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις και σε επιπτώσεις στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αναδείχθηκε άλλωστε από όλη τη συζήτηση η ανάγκη ε, μιας νέας διαθεσμικής σχέσης με την Κομισιόν, στην οποία φαίνεται ότι η Κομισιόν και δεν αναφέρομαι στο ρόλο της, της Διεύθυνσης Γεωργίας, του Επιτρόπου για θέματα Γεωργίας, αλλά του Επιτρόπου για θέματα διεθνούς εμπορίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και οι ενστάσεις μας αναφέρονται σε εκείνο ακριβώς το κομμάτι. Και στην, ε, σε ό,τι αφορά η κυρία Γέγκλη επανέφερε το ζήτημα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και στο αίτημα του, του Καναδά για την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομασία προέλευσης και ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και επί των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Καναδά, το οποίο πράγματι είναι και αυτό μια κορυφαία εμπορική δύναμη και ο Καναδάς και μας αφορά ως Επιτροπή Γεωργίας. Ο κ. Μάτο αναφέρθηκε σχέση με Περού, Κολομβία, Μερκοσούν, Σακαράνια νησιά, Μπανάνα και ε, κατανοώ το εύγλωτο ενδιαφέρον του για το θέμα της, ε, της μπανάνας. Κυρία Μαγκίνες, και αυτή στη σχέση με Μερκοσούρ και στην εισαγωγή βοήου κρέατος, αλλά και σκαυτηρίασε επίσης και η ίδια τη στάση της Κομισιόν και συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις της κυρίας Ντότς για την επιστημική ασφάλεια και την ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο σημείο 2 της έκθεσής μου, όπως επίσης και στο ε, ζήτημα της αγωγής βοήου ε, κρέατος. Θα ήθελα ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους τον κύριο Καπούλα Σάντος που μας ενημέρωσε ε, για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις χώρες Μερκοσούρ και για την επικείμενη μελέτη ε, του αντικτύπου που πρόκειται ε, να εμφυλοχωρήσει, να έλθει, ώστε να έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα για αυτό το τεράστιο ζήτημα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ε, κοινή αγοράς του Νότου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Πατράου Νέβες ε, και ιδιαίτερα ε, στις τρεις πτυχές που αναφέρθηκε στο τέλος της παρέμβασής της, δηλαδή στους δύναμους κανόνες, στην αξιολόγηση επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου και στην ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και στον ε, κύριο Λαβία, με τον οποίο μας συνδέει, βλέπετε, σχέση καλής γειτονίας και εδώ, αλλά και ως χώρες, και για ότι δεν αρκούν τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις μπανάνες, αυτά τα παραδείγματα, και έκανε και ο ίδιος έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις με το Μαρόκο και τις επιπτώσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο, στις ευρωπαϊκές χώρες. Ε, χάρηκα που άκουσα από τον κύριο Σιβένα να αναφέρεται και στο ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του γύρου της Δόχα ε, εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στη λογική του ενιαίου πακέτου, της ενιαίας δέσμευσης, ε, του ενιαίου εγχειρήματος, αυτού του single ε, undertaking, και, ε, και όπως επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω και για τα, τις αναφορές στα γεωγραφικά στοιχεία τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην άκτα και ότι είμαι πολύ χαράκουσα ότι ο κατάλογος των ε, γεωγραφικών ενδείξεων δεν είναι κλειστός κατάλογος αλλά μπορούν να προσθεθούν ε, και νέες περιπτώσεις. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα όσο γίνεται πιο γρήγορα να αντιδράσω ε, στις παρατηρήσεις πάρα πολύ δημιουργικές των συναδέλφων και θέλω να πιστεύω ότι η συνεργασία μας σε επίπεδο τροπολογιών θα είναι εξίσου ε, δημιουργική προκειμένου ε, το τελικό κείμενο, η τελική μας δουλειά ε, να βγάζει, να, να εκπέμψει μήνυμα και στο, προς, τους άλλους, προς τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά πολύ περισσότερο στο δυναμικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, που είναι οι αγρότες, οι Ευρωπαίοι της, της Υπέθρου, οι οποίοι δρούν, εργάζονται μοχτούν κάτω από αντίξωε συνθήκε σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη που είναι αυτή της οικονομικής κρίσης στην οποία ενδερχόμαστε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Γιώργο Παπαστάμκο και προχωρούμε με την ε, ημερήσια διάταξη υπενθυμίζοντας ότι οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα. Πράσινη βίβλος της Επιτροπής. Η προστασία των πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά δάση. Προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή μας είναι συναρμόδια Επιτροπή υπό την έννοια του άρθρου 30 του ε, κανονισμού με την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο Λούσια Νικουλέσκου είναι εισηγητής. Θα του δώσουμε αμέσως και τον λόγο για να μας περιγράψει την έκθεση. Θα ήθελα να προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ, γιατί μόλις κλείσαμε μια πολύ μακρά και δύσκολη συζήτηση. Με την πράσινη βίβλο της η Επιτροπή ζητά να απαντήσουμε μια σειρά ερωτημάτων που συνδέονται με τη σημερινή κατάσταση των δασών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα περισσότερα προβλήματα έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Κατά τη γνώμη μου, πράγμα που πρότεινα και συνέταξα, προσπάθησα να βρω απαντήσεις για, τα ερωτήματα που αφορούν τη δική μας αρμοδιότητα και θα σας τα παρουσιάσω εντάχει. Καταρχήν το πρόβλημα της επικουρικότητας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργήσει για να ε, εφαρμόσει και να συντονίσει τις πράξεις των κρατών μελών στον τομέα της δασικής πολιτικής. Η κλιματική αλλαγή θα έχει διαφορετικές συνέπειες ανάλογα με την κατηγορία των ευρωπαϊκών δασών. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική προετοιμασία πρέπει να προσδιορίζεται σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, να μπει, θέλω να υπογραμμιστεί στενή σχέση μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των δασών. Επίσης, να αντιμετωπιστούν τα δάση ως πηγή προσπορισμού εσόδων και να προσδιοριστεί και ο ρόλος των δασών στη γεωργική παραγωγή. Οι παραγωγικές πτυχές δεν έρχονται σε αντίθεση με την προστασία των δασών ή των άλλων ευεργετημάτων τους και θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Κατά τρίτο λόγο, στην... η θέση των δασών στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Ο τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας μεταφράζεται ιδίως στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ. Πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο δεύτερος πυλώνας ως αποτελεσματικό εργαλείο. Και μετά από το 2013 πρέπει να διατηρηθεί η στήριξη για τις δασικές καλλιέργειες, για τα καλλιεργούμενα δάση. Τα δάση είναι σημαντικός προμηθευτής δημόσιων υπηρεσιών που δεν ε, ανταμείβονται από την ε, αγορά όπως η προστασία της βιοπικιλότητας, ε, η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και η συμβολή του στο υδρογεωγραφικό δυναμικό. Γι' αυτό και τα δάση πιστεύω ότι πρέπει να έχουν πρόσθετη χρηματοδότηση, άμεση χρηματοδότηση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εφαρμογή του άρθρου 68 για τη δασική καλλιέργεια. Τα δάση μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων μας, έχουν ε, μεγάλες δυνατότητες ε, ως πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες, ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και δεν, τα, δεν τα εκμεταλλευόμαστε αρκετά. Τα δάση αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο σχολιασμό μου και τώρα θα αναμείνω τι προτάσει σα και τι τροπολογίε σα. Ο κύριο Μποβέ. Ευχαριστώ. Κυρία, Κυρία Κώστιγκερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νικολέσκου για το έργο που κάνατε. Θέλω να το χαιρετήσω ρητά ότι η εστίαση στην έκθεση βρίσκεται στο δυναμικό των δασών για την κοινωνική και όλας ε, τυχή και για την συνεισφορά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εκμετάλλευση και η προστασία των δασών αποκτούν μια πολύ σημαντική νέα σημασία. Η αρμοδιότητα σε σχέση με τα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί, εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε ιδιαίτερα τις περιφερειακές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες στα κράτη-μέλη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης πρόκειται για το θέμα ποιες είναι οι προσεγγίσεις ώστε πανευρωπαϊκά στο μέλλον να έχουμε οικολογικά μέτρα για την αηφορία στη δασοπονία που θα υιοθετούνται. Νομίζω η προσέγγιση της αηφορίας και της κάλυψης μέσω αηφόρων πηγών ενέργειας των ορυκτών καυσίμων θα δώσει απόλυτη πρόσθετη αξία σε σχέση με την κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως συνθήκες πλαισίου και για την προστασία του κλίματος και για την ενεργειακή πολιτική πιο αποτελεσματικά. Εδώ πρέπει συγκεκριμένες απαντήσεις και μέτρα να δοθούν. Η συζήτηση για την κλιματική προστασία δεν πρέπει απλά και μόνο να λαμβάνει υπόψη την προστασία του δάσους. Στόχος πρέπει να είναι η αηφορία στην χρήση και στην εκμετάλλευση των δασών. Θα ήθελα όμως ε, να καταθέσω και κάποιες τροπολογίες ως προς αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Χέκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το κείμενο. Το εκτιμώ. Από την άλλη πλευρά έχω κάποια σχόλια να κάνω. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, ποικιλότητα των διαφόρων εθνικών συστημάτων πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε ορισμένες πολύ μεγάλες, σε άρες, ο βαθμός ιδιοκτη... Ε, κρατικής ή ιδιοκτησίας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η ιδιωτική ιδιοκτησία κυριαρχεί σε μερικές χώρες, όχι μόνο για τα δάση, αλλά και για τη διαχείρισή τους. Υπάρχουν ιδιόκτητα δάση δηλαδή σε πολλές χώρες. Χρειάζεται προσαρμογή βέβαια λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία σε άλλη, στην υπόλοιπη περιβαλλοντική νομοθεσία ε, είναι διαφορετική. Εμείς την προσαρμογή τη βλέπουμε ως τη δυνατότητα των δασών μας να συνεχίσουν να παρέχουν αυτά που παράσχουν. Αποτελούν τη βάση της οικονομίας σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές και υπάρχουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα και αποτελούν και τη βάση ενός πολύ ανταγωνιστικού κλάδου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας αυτό κατά νου, νομίζω ότι τα δάση πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με αηφόρο τρόπο. Φυσικά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην διατήρηση ορισμένων περιοχών για λόγους ε, διατήρησης της βιοπικιλότητας ε, και, σε άλλες περιοχές να, έχουμε μια βιώσιμη δασοκαλλιέργεια. Νομίζω ότι πρέπει και αυτές τις δύο πτυχές να τις διατηρήσουμε σε σωστή ισορροπία. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνο η επικουρικότητα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δάση υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς, σε διαφορετικούς κανόνες από ό,τι η γεωργία. Και παρόλο εδώ είναι η καθόλου σεβαστή Επιτροπή Γεωργίας. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αγορά όσο αφορά τα δασικά ζητήματα. Νομίζω ότι σε, ότι σε πολλά μέρη της Ευρώπης έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν και να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα αλλά και να έχουμε δασοκομεία η οποία την οποία τη διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο που διατηρεί την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας. Αυτό έχει μεγάλη σχέση για μας, για την ομάδα των φιλελεύθερων. Επίσης, συμφωνώ μαζί σας ε, για την έλλειψη γνώσεων που υπάρχουν σε πολλές από τις υπηρεσίες ε, στις Βρυξέλλες. Χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις, χρειαζόμαστε τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια πλαίσια, τον ίδιο τρόπο καταγραφής και τήρησης στατιστικών στοιχείων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Επίσης χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη έρευνα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ήδη βλέπουμε στην Σουηδία, στα υψηλά βουνά ε, του Νότου, ε, βλέπουμε αλλαγές που δεν ε, τις βλέπαμε ούτε στα βιβλία της ιστορίας ούτε στη μνήμη μας. Δηλαδή το κλίμα ήδη επηρεάζει τα δάση μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τα έντομα, τις νόσους που πλήττουν τα δάση λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών. Και στην, Πορτογαλία, στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, τα δάση της Πορτογαλίας θέτουν, κρούν, θέτουν ένα θέμα συναγερμού από τις επιθέσεις των, ενστικ, ε, εντόμων. Με συγχωρείτε. Πρέπει να επιδιώξουμε μία συνένεση για την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, για την διαχείριση των δασών, για την ε, διαχείριση της καταστροφής των δασών, της αποψήλωσης, της αναδάσωσης κτλ. Χρειαζόμαστε ενεργό συνεργασία χρειαζόμαστε ένα κομβικό σημείο μέσα στην Επιτροπή όπου να μπορούν να συγκεντρώνονται όλες οι γνώσεις και πληροφορίες έτσι ώστε να έχουμε ένα κέντρο εμπειρογνωσίας αν θέλετε για όλα τα δασικά θέματα. Σήμερα το, η αρμοδιότητα αυτή είναι κερματισμένη, κατακερματισμένη και αυτό δημιουργεί χαμηλότερη ποιότητα σε διάφορους κλάδους της πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό στοιχείο, είτε αυτό αφορά τη στατιστικά στοιχεία, είτε την έρευνα, είτε ό,τι άλλο θεωρούμε ό,τι αφορά την, τα δάση, τη δασοκομεία. Επίσης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για τις αλλαγές της χρήσης γης, καλό θα ήταν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών να διευκρινιστεί η παράγραφος 3, σημείο 3. Υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις ε, της έννοιας χρήση γης ή αλλαγή της χρήσης γης και έμεση αλλαγή της χρήσης γης. Ε, η, η μία απορρέει από προτάσεις και διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι κάτι πάρα πολύ διοικητικό, πάρα πολύ γραφειοκρατικό, πάρα πολύ δυσβάσταχτο για, τους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό είμαι κατά. Δεν είμαι κατά της συζήτησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, αλλαγή χρήσης ε, των δασών υπό ευρύτερη έννοια είναι μια απαραίτητη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι για την Επιτροπή μας και για όλους όσους ενδιαφέρονται για τα δασικά ζητήματα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό στο τελικό κείμενο να προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα όρια των, ε, των δύο αυτών διαφορετικών συζητήσεων και πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Και με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό κείμενο και θα επανέλθω με τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Εκ και δίνω το λόγο τώρα για Εκεί κάτω, εκεί κάτω είναι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μετά από αυτή την επισήμαση πραγματικά θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή με ένα τρόπο συμπυκνωμένο θεμελιώδη, τα θεμελιώδη στοιχεία εμπεριέχονται εδώ. Η δική μου παρέμβαση αφορά περισσότερο την προσοχή που πρέπει να δώσουμε για την ανάπτυξη κάποιων πτυχών που θεωρώ ότι είναι σημαντικά κυρίως όταν όλοι συμφωνούμε σίγουρα, και αναφέρθηκε αυτό εδώ από την συνάδελφο Κόστιγκερ, ότι έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία κάθε μέρα τα δάση. Είναι οικονομική αξία των δασών, κοινωνική αξία, περιβαλλοντική, βιολογική και για το παιχνίδι και την αναψυχή και πρέπει έτσι να συνεχίσουμε. Θα είναι όλο και μεγαλύτερη σημασία των δασών και η υποχρέωσή μας είναι να διασφαλίσουμε την συντήρησή τους και την διασφάλισή τους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όσον αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δάση, θα έπρεπε να αναπτύξουμε μια πολιτική συμπυκνωμένη και συντονισμένη. Και γι' αυτό είμαι υπέρ μιας πολιτικής δασοπονίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ισορροπία που θα είναι σωστή και καλά μελετημένη σε σχέση με εκείνο το οποίο θα είναι κοινές ε, ε, κοινοτικές αρμοδιότητες και από την άλλη πλευρά αρμοδιότητες των κρατών μελών, κυριαρχικά τους δικαιώματα. Εδώ λοιπόν είναι η πιο δύσκολη πτυχή αυτή η ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί. Αν, αν όμως εμείς ε, δεν κάνουμε συντονισμένες δράσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δάσος ως δημόσιο αγαθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απειληθεί και μάλιστα θα απειληθεί έντονα. Και για την προστασία των δασών είναι σαφές ότι πρέπει και τα δύο σκέλη να χρησιμοποιηθούν όπως αναφέρεται στην έκθεση. Η προστασία, ένα σκέλος, και η συνιστόσα προσαρμογής από την άλλη. Προστασία και προσαρμογή λοιπόν. Όσον αφορά και τις δύο αυτές πτυχές, Πάντα πρέπει να δίνουμε προσοχή σε αυτά που είναι οι ιδιομορφίες και οι ιδιαιτερότητες των δασών, των περιοχών των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τέτοιο τρόπο ώστε να, είναι, να σεβόμαστε τη φύση, αλλά ταυτόχρονα με τις επιστημονικές γνώσεις που έχουμε πλέον σήμερα και με την επιστημονική υποστήριξη για απόκτηση περισσότερων γνώσεων να σκεφτούμε τρόπους και μορφές προσαρμογής τους ώστε να αντιδράσουμε σε αυτά τα οποία αφορούν και πλήττουν τα δάση ιδιαίτερα, τις πυρκαγιές δηλαδή, και να τις αντιμετωπίσουμε και να συνεισφέρουμε ώστε οι δράσεις για τον έλεγχο των κλιματικών αλλαγών να ενδυναμωθούν. Τελευταία πτυχή που δεν μπορώ να αγνοήσω αφορά τις δασοπυρκαγιές, τις πυρκαγιές που ο εισηγητής ανέφερε στην τελική εκ, εκ, διατύπωση του κειμένου, στην τελική έκθεση και που βιαστικά ε, αναφέρθηκε στο τελευταίο στοιχείο. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το στοιχείο θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο, να ενδυναμωθεί περισσότερο στη γραμμή εκείνων που είναι διάφορες και αλληλοδιάδοχες θέσεις που είχε υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερα η δική μας Επιτροπή ε, Γεωργίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασοπυρκαγιές είναι η απειλή, η μεγαλύτερη απειγή πιστεύω εγώ, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για την προστασία των δασών. Αφορά και πλήττει την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τα κράτη του νότου της Ευρώπης, και έτσι καθώς αφορά οι δασοπυρκαγιές αφορούν τα δάση του Νότου, αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει σε σχέση με τις δασοπυρκαγιές να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το θέμα σε σχέση με τις ευρείες συμφωνίες που έχουν ήδη συναυθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Όσλιν. Ναι, Πρόεδρε, κάποιε σύντομε παρατηρήσει μόνο, γιατί σε μεγάλο βαθμό είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση. Βρίσκω ότι η Ευρωπαϊκή Δασοκομεία και Δασοπονία πρέπει να περάσει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας σε σχέση με άλλες χώρες αφορά αυτή την πτυχή των δασών. Αλλά και για μας το θέμα αυτό μόνο στο περιθώριο, περιθωρίο έχει αντιμετωπιστεί. Σημείο 1 λοιπόν Έχουμε πολλά προβλήματα για, με τα δάση και λόγω ε, των κλιματικών αλλαγών. Και μπορούν όλα αυτά να είναι σοβαρή απειλή πολλών ε, ε, οικοσυστημάτων και δασοσυστημάτων. Πρέπει σε πολλά σημεία και μέτωπα να δράσουμε θα πρέπει να γίνει σταθερότερο το πλαίσιο, δηλαδή να γίνουν περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες και περισσότερες συμβουλευτικές δραστηριότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθεί υποστήριξη για τη σταθεροποίηση και διατήρηση των δασών. Αλλά και η πτυχή του περιβάλλοντος πρέπει να ληφθεί υπόψη στα μέτρα μας. Πολλές περιοχές ε, όσον αφορά τα δάση έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Natura 2000, στο δίκτυο Natura 2000. Μετά αγνοήσαμε όμως δυστυχώς να διασφαλίσουμε χρηματοδοτικά μέσα κονδύλια για την προώθηση προαγωγή της δασοπονίας ε, την διασφάλιση των δασών. Θα είχα την πρόταση να αναφέρουμε ότι σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει η εκμετάλλευση των δασών να αναπροσαρμοστεί, να γίνει εκμετάλλευση μεικτών δασών, κονοφόρων και φιλοβόλων. Έχουμε λάθος δέντρα σε πολλές περιοχές που έχουν φύτευθεί και που πολλές φορές ε, βρίσκονται σε λάθος σημείο για την εκμετάλλευση. Πρέπει να υπάρξει προσαρμογή αυτών των ειδών. Θα ήθελα για να τονίσω την πτυχή της δασοκομείας στην έκθεση να καταστήσουμε σαφές ότι για πολλές περιφέρειες είναι μια πολύ σημαντική ε, συνιστόσα για τη διασφάλιση της απασχόλησης, για την εργασία πολλών ανθρώπων που διασφαλίζεται έτσι από τη δασοκομεία. Και οι προαλαλήσαντες το ανέφεραν. Είχαμε μεγάλες απώλειες δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω λόγω δασοπυρκαγιών. Επανειλημμένα αλλού έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στις διαβουλεύσεις μας. Δυστυχώς έγιναν πολύ λίγα πράγματα εντωμεταξύ στο μεσοδιάστημα. Διαβάζουμε στις... το καλοκαίρι ότι καίγονται ολόκληρα δάση από τις δασοπυρκαγιές. Στη συνέχεια δεν έχουμε στοχοθετημένα μέτρα αναδάσωσης. Δεν έχουμε μακροπρόθεσμα μέτρα προστασίας αυτών των οικοσύστηματων. Αυτά πρέπει κατεπηγόντως να αποκατασταθούν και να αλλάξει η νοοτροπία και η δράση μας γιατί διαφορετικά θα έχουμε τεράστιες απώλειες δασών στην περιοχή του νότου της Ένωσης που πολύ δύσκολα μπορούν να αποκατασταθούν και να, να ζωογονηθούν. Πρέπει κατεπηγόντως να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που συχνά έχει αναφερθεί να γίνει πράξη στο τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Όστλινγκ. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο παράγραφοι χρειάζονται κάποια αποσημείωση, 4 και 5. Ιδίω η 4 που αφορά τη χρηματοδότηση. Όπου ζητάτε μια εξισορρόπηση μεταξύ δασοκομείας και γεωργίας και πιο αποτελεσματική κατανομή των κοντιλίων. Αυτό θα χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση. Και στην 14 δεν είμαι σίγουρη αν φταίει η μετάφραση ή η διατύπωση λέει υπερβολική αναδάσωση, τι εννοεί αυτό, μήπως εννοεί αποδάσωση. Μέτερ. Ο κύριος Καπούλας και Σάντος και θα πάρει πάλι τη θέση του ο Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ο εισηγητή αναφέρει στο σημείο 12 τη έκθεση του ότι θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε και να ενθαρρύνουμε τι ενώσει ιδιοκτητών αυτό είναι μια πτυχή πάρα πολύ σημαντική, τεράστια σημασία στα κράτη-μέλη, όπου ιδιωτικά δάση είναι, ουσιαστικά τα δάση είναι ιδιωτικά. 95% στη χώρα μου είναι τέτοιου είδους ιδιωτικές ζώνες ε, δασών και όπου σε πολλές, σε πολλές ζώνες έχουμε μικρές ιδιοκτησίες. Οποιαδήποτε πολιτική συντονισμού για τα δάση, η καλύτερη δράση πρόληψης για τα δάση δεν έχει την μεγάλη διάσταση συντονισμού μεγάλων δασών. Και τώρα θα πρέπει εδώ να δούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιου είδους μεγάλη, μεγάλο συντονισμός όταν είναι μικροϊδιοκτησίες. Θα ήθελα λοιπόν να, να πω στον κύριο εισηγητή ότι θα ήθελα να εντάξει με έναν τρόπο πιο σαφή και πιο αποσαφηνισμένο το ότι πρέπει περισσότερο από το να ενθαρρύνουμε να εντάξουμε σε ένα πλαίσιο. Θα μπορούσε το άρθρο 68 να είναι η βάση για αυτή την δράση. Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί σας κύριε Ισηγητά να βελτιώσουμε το σημείο 10 και το σημείο 12 στην έκθεσή σας ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη αυτές οι μεγάλες ανησυχίες στις οποίες αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. E Ευχαριστούμε Λουίς και θα λάβει στην συνέχεια τον λόγο η πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Χάμελ παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Yes. Thank, thank you. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα αυτό στη σύνταξη της Πράσινης Βίβλου είχαμε συνειδητοποιήσει ιδιαίτερα τις διαφορετικές ε, αρμοδιότητες και τους διάφορους τομείς διαφορετικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δάση και καταστήσαμε σαφές δύο πράγματα. Καταστήσαμε σαφή. Πρώτα απ' όλα το θέμα της επικουρικότητας. Αυτό είναι ένα έγγραφο που θέλει να ξεκινήσει μια συζήτηση, αναγνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν κλιματικές αλλαγές και μετά στη συνέχεια λέγοντας εντάξει λοιπόν, τούτου λεχθέντος πώς μπορεί η ευρωπαϊκή πολιτική να αναπτυχθεί και να μετεξελιχθεί ώστε να συνεισφέρει στις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Ήταν απόλυτα σαφές σε αυτόν τον τομέα που βρίσκονται λοιπόν οι ευθύνε και οι αρμοδιότητες και το ότι κοινοτικές προσπάθειες είναι προσπάθειες πρόσθετης αξίας ως δράσης και η δεύτερη πτυχή που νομίζω έχει τεράστια σημασία υπό το δικό μας πρίσμα είναι ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλο το έγγραφο, στα παραγωγικά στοιχεία, στα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και στο περιβάλλον και όλες αυτές τις συνιστώσεις συνολικά. Διότι απόλυτα γνωρίζαμε και είχαμε συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να δράσουμε χωρίς το ένα στοιχείο ή χωρίς το άλλο. Η δυσκολία τώρα ποια είναι η δυσκολία και η πρόκληση είναι και όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό και γι' αυτό η συνεισφορά αυτή τη κοινοβουλευτική σα επιτροπή και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία για μα. Η δυσκολία τώρα βρίσκεται στο να συμφιλιώσουμε και να συγκεράσουμε διαφορετικά συμφέροντα όσον αφορά την προστασία των δασών και στο να συμφιλιώσουμε και συγκεράσουμε τα την ίδια τα στοιχεία αυτά ως προς τη συνθήκη στο εύρος κατά το οποίο μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και συνδρομή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινότητα μέσω των διαθροτικών ταμείων, του Ταμείου Ανάπτυξης της Υπέθρου κτλ. Προ το συμφέρον πάντα όπως και το ζητούσε η κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και με χαρά βλέπουμε ότι τονίστηκε από τα μέλη της επιτροπής σα η ανάγκη για την πληροφόρηση και ενημέρωση. Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριακών στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση των δασών. Πολλά από αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία βρίσκονται όχι σε κάποιο ε, σε κάποια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες δεδομένων όσο αυτά τα κράτη-μέλη και ειδικά για τα δάση τέτοιου είδους βάσεις δεδομένων. Στρεφόμαστε προς τα κράτη-μέλη να δουν και να αντιληφθούν γιατί πρέπει να μοιραστούμε αυτά τα στοιχεία και ποια στοιχεία πρέπει να μας διαβιβάζουν. Αναφέρθηκε το ότι έχουμε δάση σε μια περιοχή που έχουν ιδιομορφίες και είναι διαφορετική η δομή τους από τη δάση σε άλλες περιοχές. Και αυτό το αναγνωρίζουμε. Δεν προσπαθούμε με κανένα τρόπο να βρούμε εύκολες ισοπεδωτικές, παγκοσμιοποιημένες ε, ισοπεδωτικές λύσεις. Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Με τέτοιο τρόπο να συνεργαστούμε ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες, πληροφοριακά στοιχεία που έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κράτη-μέλη τα ίδια, να χρησιμοποιήσουμε και εκμεταλλευτούμε αυτά τα στοιχεία εμείς οι ίδιοι, αυτά που μπορούν να προσαρμόσουν τις δασο, δασικές πολιτικές ώστε να είμαστε πιο παραγωγικοί κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τη διαχείριση των δασών. Το Συμβούλιο αντιμετωπίζοντας αντιμετωπίζοντας την λευκή βίβλο όσον αφορά προσαρμογές, προσαρμογές πέρυσι νομίζω που έγινε αυτό, με ιδιαίτερη προσοχή έλαβε υπόψη την έκθεση του 2009 της, ε, ε, των ενώσεων ερευνών ε, για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αναφέρθηκε ότι ο προηγούμενος αιώνας επηρέασε πολύ σημαντικά τα, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δάση και υπάρχει κίνδυνος εδώ λόγω και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα να απολεστούν τα δάση εκτός αν μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτά τα συμφέροντα ο άνθρακα το διοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα επιδεινώνει τις κλιματικές αλλαγές και αυτό απειλεί τα δάση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πρόκληση και είναι προς το συμφέρον του τομέα να μπορέσει το δάσος να λειτουργεί ως αφομοιωτή του ε, διοξιδίου του άνθρακα και να μην ε, ε, μέσω αυξημένων θερμοκρασιών και ε, διοξιδίου του άνθρακα που εκλείται στην ατμόσφαιρα αντί να αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος να γίνει μέρος του προβλήματος του ίδιου. Πρέπει λοιπόν να προστατευτεί το δάσος και έτσι σε σχέση με τη δράση του Κοινοβουλίου και τις γνωμοδοτήσεις των εμπλεκομένων ε, ενδιαφερομένων κύκλων και του Κοινοβουλίου έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας θα μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και συνεργαζόμενοι σε πολύ στενό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους, να προσπαθήσουμε να βρούμε μία οδό με την οποία μπορεί να συνεισφέρει καλύτερα η κοινότητα στην προστασία των δασών για όλους τους λόγους που προανέφερα και σεβόμενοι πάντα απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που σχολίασαν ή έκαναν συστάσεις. Όπως είπα από την αρχή, ε, εργαστήκαμε μέσω με τη συνεργασία, σε συνεργασία με την Κομισιόν και πολλά από αυτά που είπατε που είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα θα αναφέρονται στην τελική έκθεση που θα γράψει η αρμόδια Επιτροπή ως προς την ουσία, η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα, το συζητήσουμε, θα την συζητήσουμε την έκθεση μετά από τη δημόσια διαβούλευση που θα γίνει την ακρόαση δηλαδή για τη δασοκομεία και τη γεωργία. Θα προσπαθήσω τώρα μία-μία να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Η βιώσιμη διαχείριση των δασών είναι πολύ σημαντική πτυχή του θέμου του προβλήματος. Κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Είμαι βέβαιος ότι αυτά θα είναι με τμήμα της έκθεσης της Αρμόδιας Επιτροπής. Εγώ το έθιξα στα πλαίσια των δικαιοδοσιών της δικής μας Επιτροπής και νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχουμε να πούμε είναι το δάσος ως βασική μονάδα της ε, υπεθρίου μονάδος. Ξέρω αυτά που είπε η κυρία Πατράου για τα δάση, τις ανησυχίες της και απαντώ έτσι και στην κυρία Μαγκίνες ότι είναι πρόβλημα διατύπωσης γλωσσικός και εγώ στη δική μου μετάφραση αυτό το πρόβλημα βλέπω. Τώρα για τον κύριο Καπούλα Σάντος. Μιλήσαμε για μακρού σήμερα για τις διάφορες ε, καταστάσεις που ισχύουν στα διάφορα δάση της Ένωσης Στη Ρουμανία έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αποδάσωσης ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Επίσης οι ιδιοκτησίες διαφέρουν πολύ. Χρειάζεται λοιπόν και μια σωστή διαχείριση μεγάλων δασοκομικών, δασικών εκτάσεων και θα ήθελα η κατάσταση να είναι παντού βιώσιμη, όχι μόνο σε μία χώρα μέλος, σε όλες. Πολλά από τα θέματα που εφήγησαν θα αναφέρονται στην έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής. μίλησα για συνέργεια μεταξύ γεωργίας και δασοκομείας. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο αυτό που λέω, αλλά κατά τα υπόλοιπα είμαι σίγουρος ότι όλα όσα είπατε, το ξαναλέω για εκατοστή φορά, θα βρεθούν στην τελική ομοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην τελική έκθεση εκείνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. κύριε Νικουλέσκου. Συνεχίζουμε τώρα. Τελευταίο σημείο για σήμερα, το 7. Τροποποίηση της οδηγίας 2018 για τη δυνατότητα των χωρών μελών να μειώσουν ή να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και φυτών στο έδαφος των ιδιαίτερα λεπτό σημείο και γι' αυτό η συζήτηση θα είναι σημαντική. Τίθενται πολλά ερωτήματα και απορίες όντως ως προς τον κίνδυνο επανεθνικοποίησης της αγροτικής πολιτικής. Ας μην προτρέχω όμως, είμαι βέβαιος, επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση θα είναι πολύ ενδιαφερούσα μετά από την αρχική εισήγηση του Γεωργίου Λάιον Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να υπάρξει συνένεση εδώ μέσα με αυτό το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Θα αναφέρω γρήγορα γρήγορα ορισμένα από τα θέματα που τίθενται μετά από την πρόταση της Κομισιόν και θα ήθελα σήμερα να ακούσω απόψεις των συναδέλφων και ως για το περιεχόμενο αλλά και για τη γενικότερη πολιτική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως Επιτροπή. Ορισμένα γεγονότα πρώτα. 14 εκατομμύρια γεωργοί το 2009 άρχισαν να καλλιεργούν ε, βιοτεχνικά και πολύ λιγότεροι από τρίτες χώρες. Αύξηση 7% σε σύγκριση με το 8%. Βέβαια μόνο δύο βιοτεχνικά είδη έχουν ε, εγκριθεί και περιμένουν ακόμη 17 πολλά επί πολλά χρόνια. 94.800 εκτάρια καλλιεργήθηκαν έτσι, που είναι λιγότερα από το 2008. Και η Ισπανία είναι η μεγαλύτερη χώρα, είναι η χώρα που καλλιεργεί τα περισσότερα τέτοια τροποποιημένα. Αυτά ως προς το φόντο. Και τώρα να δούμε τη συγκεκριμένη πρόταση, όχι τα υπέρ και τα κατά των τροποποιημένων, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Και ιδιαίτερα την τροπολογία να συζητήσουμε προ του Επιτρόπου Βάλλη. Λέει ως δικαιολόγηση της πρότασής του ότι θα χρειάζεται μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία διοδότησης και ότι τα κράτη-μέλη, τα κράτη λέγω μέλη, δεν θα μπορούν να κρύβονται όταν θέλουν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια κάποιου είδους. Και συνεχίζει η Κομισιόν εξηγώντας την τροπολογία αυτή στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η αδειοδότηση και να ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες όπως οι ρήτρε ασφαλείας που επικαλούνται πολλές φορές τα κράτη-μέλη εφόσον όμω βασίζεται, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον βασίζεται σε ατράνταχτα επιστημονικά στοιχεία. Πιστεύουν λοιπόν ότι έτσι θα μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος και για την ΕΦΣΑ και για την Κομισιόν. Η συνθήκη βέβαια προβλέπει ότι η καλλιέργεια των τροποποιημένων φυτών δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο αν υπάρχουν οι απαραίτητες υγειονομικές και περιβαλλοντολογικές εγγυήσεις. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή νομική και Τέλος, λέει η Επιτροπή ότι έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους ενδιαφερόμενους, για τους όσους καλλιεργούν τροποποιημένα, για όσους καλλιεργούν φυσικά, για τους κτηνοτρόφους κλπ. Και ίσως να αυξήσει κιόλας και την προβλεψιμότητα, λέει, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έτσι δικαιολογεί η Κομισιόν την πρότασή της. Και μερικά από αυτά που λέει είναι πενετά και Πενετέα. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι το 12 θα γίνει μια αναθεώρηση γενικότερα της νομοθεσίας που αφορά τις αδειοδοτήσεις για καλλιέργεια τροποποιημένων. Τους κανονισμούς και τα λοιπά σε δυο περίπου χρόνια λοιπόν. Όταν άρχισα να εξετάζω το θέμα αναρωτήθηκα καταρχάς εάν εμείς ως Επιτροπή δεχόμαστε την ίδια την αρχή της πρότασης, δηλαδή επανεθνικοποίηση των αποφάσεων για την καλλιέργεια ημίτροποποιημένων. Και η δεύτερη αρχή που κρύβεται από πίσω είναι αν τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα ή όχι με βάση επιστημονικά στοιχεία να εφαρμόσουν απαγόρευση. Νομίζω ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα και εγώ νομίζω ότι η βάση όλων αυτών, δηλαδή η επιστημονική γνώση που προτείνεται σαν βάση, για την ασφάλεια ημία αυτών των προϊόντων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν δει κανεί πόσες νέες τεχνολογίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, η νανοτεχνολογία και όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις. Καταρχήν λοιπόν δεχόμαστε ή όχι την αρχή της επανεθνικοποίησης, δεύτερον δεχόμαστε ή όχι την αρχή ότι μπορούν να υπάρξουν και λόγοι άλλοι μη επιστημονικοί για την απαγόρευση των νέων αυτών τεχνολογιών. Δεύτερο θέμα. Συμμεριζόμαστε ή όχι τις ανησυχίες ορισμένων εταιριών και γεωργών ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέες αυτές αποφάσεις και καλλιέργειες στην αγορά, στην ενιαία αγορά αν επιβληθούν τέτοιες μεμονωμένες απαγορεύσεις. Η Κομισιόν δέχεται ότι υπάρχουν εδώ προβλήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Αν δεχτεί κανείς λοιπόν αυτές τις αρχές, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι δεχόμαστε ή όχι τα κριτήρια με τα οποία πρέπει τα κράτη-μέλη να δικαιολογούν τις σχετικές τους αποφάσεις τι λόγο μπορεί να δώσει ένα κράτος μέλος εκτός από επιστημονικούς και περιβαλλοντολογικούς. Επιβάλλεται ο σεβασμός των συνθήκων και των κανόνων του ΠΟΕ. Τι μένει λοιπόν ως λόγος, ηθική, δεοντολογική λόγη, δημοψήφισμα όπου ένας λαός αρνείται μια καλλιέργεια και τότε απαγορεύεται και αυτό θα ήταν πρωτοφανές. Επόμενο ερώτημα. Τι προσθέτει αυτή η πρόταση. Αν η Κομισιόν δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα επιταχυνθεί έτσι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα καταλήξουμε πάλι σε πάγωμα στο Συμβούλιο, τι αξία έχει αυτό, τι προσφέρει η πρόταση. Ξέρω ότι μερικές χώρες μέλη ζήτησαν τέτοιες προτάσεις, αλλά αν δεν λύνεται το πρόβλημα του παγώματος στο Συμβούλιο, τι αξία έχει. Θα καθησυχάσουν έτσι τις ανησυχίες ορισμένων χωρών μελών για τις απαγορεύσεις που έχουν εφαρμόσει ή θέλουν να εφαρμόσουν απαγορεύσεις. Θα σταματήσει τα κράτη-μέλη από τη χρησιμοποίηση της ρήτρας ασφαλείας ή απλώς θα δώσει το πολιτικό μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να έχουν εκείνα την ευθύνη. Και αν ναι, το δεχόμαστε αυτό το παιχνίδι. Πώς να εγγυηθούμε ότι αυτή η πρόταση θα εγγυάται την ελευθερία όλων των γεωργών ως προς το τι πρέπει και θέλουν να καλλιεργήσουν και μάλιστα με τρόπο συγκρίσιμο για τις υπόλοιπες χώρες εφόσον υπάρχει πανενωσιακός ανταγωνισμός και διεθνής. Τι όρια προβλέπονται για τα γενετικώς τροποποιημένα τρία, γάμα ταφ 3. Τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στην ενιαία αγορά αν είναι πολλοί και πολλαπλοί οι ορισμοί του τι είναι γενετικός τροποποιημένος οργανισμός. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε για τη νομική βεβαιότητα που μπορεί να έχει μια τέτοια πρόταση. Γιατί εγώ νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί οποιαδήποτε απόφαση κράτους μέλους αν δεν είναι 100% σίγουροι και θα χρειάζεται για κάθε περίπτωση νομική γνωμοδότηση. Ο συνάδελφός μου, Κόραν Λεπάζ, η συνάδελφός μου Κορίν Λεπάζ που είναι μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος ζήτησε γνωμοδότηση από τις, κοινοβουλευτικές, από τις αρχές του Κοινοβουλίου. Θα έχουμε λοιπόν τουλάχιστον δύο νομικές γνωμοδοτήσεις τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να πει ότι δύο χρωματοδοτήσεις είναι καλύτερες από μία, αλλά τέλος πάντων. Αν υπάρχει νομική βεβαιότητα λοιπόν για τις προτάσεις αυτές. Αυτό, αυτή η πρόταση μάλλον αφηνήσει κάπως τα πράγματα ή όχι. Είπα ότι υπάρχουν ήδη προβλήματα με τον ορισμό. Μπορεί να καταλήξουμε σε 27 διαφορετικούς ορισμούς περί του τι είναι γενετικός τροποποιημένος οργανισμός 3. Γιατί σύμφωνα με τους νέους κανόνες τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν και τι θα συγκαλλιεργούν μαζί με τους γενετικούς τροποποιημένους. Συμφωνούμε ότι έτσι χρειάζεται να γίνει ή να ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για διαφορετικές ερμηνείες και παρερμηνείες. Και τελικό ερώτημα που είναι πολιτικό και δεν αφορά την ίδια την πρόταση. Τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Επιτροπή μας. Αν αποφασίσουμε ότι δεν μας αρέσει αυτή η πρόταση και την απορρίπτουμε, την αναπέμπουμε στην Κομισιόν. Τη θεωρούμε μη ρεαλιστική, ασαφή, με αναπάντητα ερωτήματα, ενώ το περιβάλλον λέει όχι εμάς μας αρέσει, είναι πολύ καλή και την προωθούμε, τότε, τότε βγάζουμε τον εαυτό μας, θέτουμε τον εαυτό μας εκτός του παιχνιδιού. Και η επίτυχε όχι τότε τι θα κάνει. Δεν έχουμε πια καμιά δυνατότητα να ξαναμπούμε στο παιχνίδι εκτός αν το κάνουμε πια ως άτομα. Αλλά αυτό νομίζω θα ήταν λυπηρό να αποσυρθούμε. Αν και βρίσκομαι στον πειρασμό να απορρίψω την πρόταση, αλλά πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η γενικότερη στρατηγική μας πριν πάρουμε τέτοια απόφαση. Εγώ και η Κορίν Λεπάζ ζητήσαμε και περισσότερο χρόνο, διότι υπάρχουν τόσο πολλά αναπάντητα ερατήματα και τόσο πολλές δυνατότητες να διαστρεβλωθούν τα πράγματα που χρειάζεται χρόνος για να το συζητήσουμε, να το καταλάβουμε όπως πρέπει πριν καταλήξουμε. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που έχουμε είναι, ίσως η γραμματεία μπορεί να με διορθώσει, κατάθεση της έκθεσής μου 10 Ιανουαρίου. Έχουμε ήδη 8 με 9 εβδομάδες για να προσπαθήσουμε να βρούμε ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Προσπάθησα να είμαι συνοπτικός. Δεν σας έδωσα πολλές απαντήσεις αλλά πολλές ερωτήσεις. Αλλά έτσι μ' αρέσει να δουλεύω με ερωτήσεις. Θα συναντηθώ με τους Κιώδης σύντομα το Νοέμβριο στο Στρασβούργο και Ελπίζω εκεί να αποσαφινιστούν κάπως τα ερωτήματα αυτά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας Πρόεδρε και προσδοκώ τις απόψεις των συναδέλφων. Πολύ καλά, Τζόρτζ. Νομίζω ότι τα έθεσες όλα πολύ σωστά και με σοβαρό τρόπο. Νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί τώρα να λάβει χώρα για να εκφραστούν οι διάφορες απόψεις. Έχουν εγγραφεί πολλοί για να λάβουν το λόγο. Αν θα είμαστε σύντομοι θα κλείσουμε σήμερα, Αλλιώ θα συνεχίσουμε και αύριο. Ο Μάρτιν έχει καταρχήν το λόγο. Μάλιστα. Τα σωστά ερωτήματα διατυπώθηκαν βέβαια. Αλλά άμα τα δει κανεί πιο κοντά αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγονται όλο και περισσότερα ερωτήματα η ομάδα μας ευθύς εξ αρχής είχε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία διατύπωσε. Τώρα μπορεί να τεθεί το ερώτημα, ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση αυτή να απεμπολίσει τις ευθύνες της σε αυτό το τομέα και να αποσυρθεί από αυτό το σκηνικό. Μπορεί να διατυπωθεί αυτό το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, θεμελιώδη ερωτήματα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο και να συζητηθούν. Σημείο 1. Ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε να εφαρμοστούν αυτά που το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ζητάει για την αδειοδότηση να ξανασκεφτούμε αρκετά πράγματα. Και αυτό δεν σε αυτό δεν ασκήθηκε ανέξοδα κριτική και αποδείχθηκε ότι πρέπει να υπάρξουν επικρίσεις και το σύνολο αυτού του θέματος πρέπει ξανά να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρκετές αρχές που γενικά είναι δεσμευτικές. Έχουμε την αρχή της συνύπαρξης, δηλαδή όλες οι μορφές γεωργικών ε, ε, ε, σπόρων έχουν τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει εδώ να δούμε ίδιοι κανόνες συνύπαρξης προϊόντων και σπόρων να υπάρχουν στην Ευρώπη. Και θα πρέπει εδώ να μην ε, υπονομευτεί αυτή η αρχή και να τεθεί το ε, θέμα των γενετικά τροποποιημένων σπόρων στο προσκήνιο. Και αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα με την νομοθεσία στην Αυστρία και σε άλλες χώρες όπου ήδη τώρα είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο για κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς, ε, να περιοριστεί η χρήση της ε, γενετικά τροποποιημένης δράσης. Και αν αυτό, αυτή την αρχή της συνύπαρξης το την θέτουμε στο προσκήνιο, τότε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ζητήσουμε να διασφαλίζει αυτά τα θέματα και τίθενται ερωτήματα εδώ. Έχουμε μια κοινή εσωτερική αγορά. Πώς θέλουμε μέσα στην Ευρώπη τελικά να εφαρμοστούν όλα αυτά και να ελέγχουμε όπως πρέπει αυτές τις προϋποθέσεις και όρους. Έχουμε το πρόβλημα των σπόρων, όπου ήδη έχουμε σήμερα ένα πρόβλημα, πράγμα το οποίο θα εντείνει το θέμα της ασφάλειας όταν θα έχουμε από τη μία πλευρά γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και από την άλλη μεριά θέλουμε να τις περιορίσουμε. Και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και τα θέματα των κανονισμών και κανόνων του ΠΟΕ και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και οι ε, ε, ε, Υπουργοί Γεωργίας και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο πρέπει να αποσαφηνίσουν αυτά τα πράγματα. Πράγματα που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. Πώς θα, έχ, θα συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη με αυτούς τους κανονισμούς και κανόνες του ΠΟΕ ή θα παραβιάζονται αυτοί. Και να θέσω και το ερώτημα ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον. Θέλουμε διεξοδικά να συζητήσουμε για αυτή την πρόταση λοιπόν. Θέλουμε αυτό το νομοθέτημα όχι μόνο σε δύο-τρία σημεία να το εξετάσουμε σε βάθος, αλλά σφαιρικά να το δούμε ολοκληρωμένα σε όλες τις συνιστώσεις του. Και πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρισκόμαστε σε περίοδο συναπόφαση, στην εποχή τη συναπόφαση και στα θέματα γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών θέλουμε να έχουμε ιδιαίτερο λόγο που θα αρθρώσουμε και σε βάθο να ασχοληθούμε με αυτά. Και για να μην τεθούμε υποπίεση χρόνου τώρα, πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται και μια και έχουμε και θέματα αδειοδότησης. Σε αυτό πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν απελευθερώνονται τέτοιου είδους καλλιέργειες πρέπει σε βάθος να εξετάσουμε τα πράγματα. Κυρίαρχα και σε βάθος να δούμε. Αν θα καταλήξουμε σε μια ενιαία λύση το αμφιβάλλω. Αλλά όλα τα στοιχεία θα πρέπει να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Bene, grazie Martin. Ευχαριστώ Μάρτιν, ο Ζωζέ Μποβέ και μετά ο κύριος Νικουλέσκου. Ναι. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή απαιτεί καταρχήν να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το, Υπουργείο, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το, την περασμένη εβδομάδα απέριψαν, και τα δύο συμβούλια απέρριψαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπαν ότι οι προτάσεις αυτές σήμερα εμφανίζονται πολύ πρόωρα σε σχέση με τα θέματα που είχε θίξει η Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε αυτά τα, αυτό το πλαίσιο, αυτά τα συμφραζόμενα. Το Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος είχε ζητήσει μία παρουσίαση της αξιολόγησης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Ομόφωνα οι Υπουργοί Περιβάλλοντας είχαν κάνει, το είχαν ζητήσει αυτό το Δεκέμβριο του 2008. Αυτό που έκανε το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα ήταν να πει «Δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει ε, να προσθέσουμε ένα άρθρο στην ε, Οδηγία 2008 χωρίς να έχουμε κάνει την προκαταρκτική δουλειά». Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ήδη από το 2008 είχε θέσει την αρχή της αξιολόγησης. Τι, θα πει αξιολόγηση. Πρόκειται για μοριακή βιολογία, πρόκειται για το περιβάλλον, ε, τα δεοντολογικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά. όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο της ε, επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. 2008 λοιπόν είχε ζητηθεί όλες αυτές οι παράμετροι να ληφθούν υπόψη. Δεύτερον, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διαφάνεια για την πραγματικότητα. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να επανέλθω στα τελευταία γεγονότα, στις τελευταίες εβδομάδες, να δούμε μόνο τι έγινε την Πέμπτη. Είχαμε το Συνδικητικό Συμβούλιο ε, και με την παρέτηση. Είχαμε το Συμβούλιο της ΕΦΣΑ, παρέτηση. Είχαμε το, αποτέλεσμα, ε, είχαμε το αποτέλεσμα των πιέσεων και του λόμπι που είχε ασκηθεί. Κλείνω αυτή την παράνθεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας λοιπόν. Έχω να πω στην, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την πρότασή σας από τη στιγμή που δεν κάνετε αυτό που σας ζητά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, ο κύριος Λάιον νομίζω είπε πράγματα θεμελιωμένα και βάσιμα. Καταρχήν για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τα σύνορα ε, και στα οικονομικά αλλά και στη ρήπανση. Έτσι θέλουμε, αλλά οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί πώς, πώς θα γίνει να εμποδιστούν να <laughs> περάσουν τα σύνορα. Αυτό δεν έχει νόημα. Είναι σαν, το σύννεφ, σαν τον νεφός του Τσέρνομπιλ, το οποίο έφτασε και στη Γαλλία. Δεν έχει λοιπόν νόημα αυτό. Μετά έχουμε το πρόβλημα της τρέβλωσης του ανταγωνισμού, κεντρικό ζήτημα. Ποια είναι η κατάσταση στη βιολογική γεωργία μιας χώρας που επιτρέπει τις γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς έναντι μιας χώρας που απαγορεύει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού εδώ. Είναι ούτε θέμα μόνο εσωτερικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο George Lyon είπε για το θέμα του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, και τελικά τι θα υπερισχύσει, το, το, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών. Η απαγόρευση ε, η απαγόρευση το να μπορούν τα κράτη να κάνουν αυτό που θέλουν δεν στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία αλλά σε οικονομικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν γίνεται. Έχουμε δει τις συνέπειες. Έχουμε δει την, τον διασκορπισμό την, της μάχης κατά των γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στο παγκόσμιο, στο διεθνές εμπόριο. Πρέπει να έχουμε αυστηρούς κανόνες. Είδαμε Είδαμε τι έγινε και με τους κανόνες για το παγκόσμιο εμπόριο. Πρέπει να εμφανιστούμε ενωμένοι και νομίζω ότι η πρόταση αυτή έρχεται σε, καλή, σε κακή ώρα, πρόωρα εμφανίζεται και πολύ κακοδιατυπωμένη είναι, κακοκατασκευασμένη. Η πρόταση των πρασίνων είναι ξεκάθαρη. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο, Νικουλέσκου, πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι εδώ έχουμε μπροστά μας μια πολύ έντονη συζήτηση. Υπάρχουν διαφωνίες όχι μόνο μεταξύ χωρών μελών αλλά και πολιτικών ομάδων αλλά και μέσα σε κάθε χώρα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις ακόμα και μεταξύ μελών της ίδιας κυβέρνησης όπως στη Ρουμανία που ο Υπουργό Γεωργίας έχει διαφορετική άποψη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να αναμείνουμε μια πολύ παθιασμένη συζήτηση. Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο απέρριψε όντω την πρόταση αυτή και αυτό δείχνει ότι δεν θέλει να δεχτεί την να αναλάβει την ευθύνη μιας απόφασης. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο Λάιον, τα ερωτήματά του είναι σωστά και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις τους. Χρειαζόμαστε πολύ πιο σαφή στοιχεία και εγώ ο ίδιος, και εγώ ο ίδιος λέγω, πρέπει να σας πω ότι η απόφαση των χωρών μελών, οι αποφάσεις των χωρών μελών πρέπει να σέβονται τη συνθήκη. Το λέει η Κομισιόν αυτό. Και άρα και την ομολογία του δικαστηρίου που ε, δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Νίκο ο Στέφανος Λεφόρ. θα ήθελα να σας πω το εξή, ο Γιώργος Λάιον έκανε μια παρουσίαση που έδειξε πόσο δύσκολο είναι, Γεώργιος Λάιον, πόσο δύσκολο είναι να αποφασίσει και ξέρουμε ότι ο Γεώργιος συνήθως όπως για την αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι πολύ σαφής. Λοιπόν, με δύο τρόπους μπορούμε να το δούμε. Ο πιο εύκολος είναι να πούμε η Κομισιόν κάνει μια πρόταση που δεν ισχύει, την απορρίπτουμε, την πετάμε και αποφεύγουμε να το συζητήσουμε. Και έτσι ο καθένας κρατάει τις θέσεις του, η μένη είναι τελείως κατά των γενετικών τροποποιημένων, η άλλη υπέρ. Και θα περιμένουμε αιωνίως να κάνει ο χρόνος το έργο του μόνος του. Και καθώς υπάρχουν υπέρ και κατά σε όλες τις χώρες, ακόμη και στην ίδια κυβέρνηση, όπως είπατε για τη Ρουμανία, βλέπουμε ότι δεν θα προχωρήσει η συζήτηση. Και η ευθύνη, η πολιτική ευθύνη ενός κοινοβουλίου είναι να προχωράει τα πράγματα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Να, καλά το είπανε πριν. Είναι σε ποιες συνθήκες θα δεχτούμε στην Ευρώπη την συγκατοίκηση, τη συνύπαρξη γενετικός τροποποιημένων και μη τροποποιημένων οργανισμών και υπό ποιε συνθήκες θα μπορούσε να οργανωθεί η συνύπαρξη. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό πρέπει να βρούμε ως απάντηση. Και βέβαια αυτά που είπε η Κομισιόν είναι ότι επιτρέπονται γενετικώς εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δεν μπορεί κανείς να τους βρει για να απαγορευτούν. Αυτό λέει περίπου. Τι πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν. Τι πρέπει να σκεφτούμε. Τέσσερα πράγματα κάτι με τέσσερα. Την υγεία, τα υγειονομικά, το περιβάλλον και με βάση την εμπειρία της μαζικής χρήσης τροποποιημένων στις ΗΠΑ υπάρχουν προβλήματα για τις φορές. Ξέρω ότι υπάρχει ένα φυτό που λέγεται αμαράντα του Πάλμερ που κανείς δεν ξέρει πώς να απαλλαγεί από αυτήν σήμερα. Λοιπόν το θέμα του περιβάλλοντος τίθεται, υπάρχει. Χρειάζεται εδώ εμπειρογνωμοσύνη. Το οικονομικό. Δεν το λέμε ποτέ αυτό. Υπάρχουν ή όχι οικονομικά συμφέροντα για τη χρήση των γενετικών. Κανείς δεν το λέει. Ε, και καμία. Αν υπάρχουν συμφέροντα να τα δούμε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι καν ενδιαφέρον οικονομικά να καλλιεργούνται τα γενετικά. Και τέταρτο, υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις στη χρήση των γενετικών τροποποιημένων. Όπως είχαμε πει για τα παρασιτοκτόνα, ζυζανιοκτόνα που θέλαμε να τα βοηθήσουμε αλλά δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Αλλά εδώ υπάρχει εναλλακτική που να είναι οικονομικά βιώσιμη βέβαια. Αυτά είναι τα τέσσερα ερωτήματα επί των οποίων πρέπει να βρούμε απάντηση. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό θα χρειαστεί χρόνος. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Η Επιτροπή Γεωργίας δεν μπορεί να αποφασίσει αν δεν κάνει πρώτα επαφές με την επαφή περιβάλλοντος. Και προτείνω να οργανωθούν τέτοιες επαφές μεταξύ Προέδρου της Επιτροπής μας, Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος, σκιωδών, για να υπάρξει μια, η λήψη μιας στρατηγικής απόφασης. Δεχόμαστε ή όχι να συζητηθεί το θέμα για να βρεθεί λύση ή μήπω λέμε απλώς τα αφήνουμε όλα αυτά και θα δούμε τι θα αντιπροτείνει η Κομισιόν. Η Κομισιόν τι κάνει επειδή την πιέζει το Συμβούλιο, προσπαθεί να προτείνει κάποια λύση που δεν την δεσμεύει. Και αφού δεν δεσμεύεται ούτε το Συμβούλιο, κανεί δεν προτείνει λύση. Και παραμένουν τα πράγματα όπω είχαν και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι η συνύπαρξη δεν είναι καλό πράγμα έτσι όπως είναι σήμερα. Ούτε για τους γεωργούς, του βιολογικού ούτε για του υπόλοιπου. Πρέπει να έχουμε μια απάντηση, μια απόφαση. Εγώ προτείνω λοιπόν μετά από αυτά που είπε ο Γεώργιος να γίνει μια συνάντηση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να γίνει μια αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα δούμε τα πράγματα στρατηγικά και αφού γίνει αυτή η αποτίμηση τότε να έχουμε τα... τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Αυτά προτείνω μετά από αυτά που είπε ο Γεώργιος. Ευχαριστώ Στέφανο. Οι επαφές με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, βρίσκονται ήδη εν εξελίξη. Νομίζω ότι κανείς δεν ε, είναι αντίθετος με τη συμμετοχή του εισηγητή μας, του George Lyon, ο οποίος θα μπορέσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο από μια απλή αναφορά γνώμης να συμμετέχει στις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες μιας μεγαλύτερης συνεργασίας, αλλά πάντως δεν μπορούμε να αποσιάσουμε από τη συζήτηση, γιατί ακόμα και αν υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία κατά αυτής της πρότασης της Επιτροπής, όπω το φαντάζομαι, εμεί παρόλα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, πρέπει να, να δηλώσουμε ποια είναι η θέση μας. Και αν απορριφθεί η πρόταση κάποια στιγμή, τι να κάνουμε. Δεν μας απαγορεύει αυτό να δηλώσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε αντίθεση με τον Ρουμάνο συνάδελφο δεν έχω το πρόβλημα διαφωνίας μεταξύ γενετικά τροποποιημένων τέτοιων καλλιεργιών από τη χώρα μας και σαν μία από τη χώρα που απεφάσισε το, ε, η αρχή της αυτοδιάθεσης να ισχύει. Παρότι σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής που έχουμε μπροστά μας, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες δημιουργούνται πολύ περισσότερα ερωτήματα από ό,τι δίνονται απαντήσεις και είναι απαραίτητο πιστεύω συγκεκριμένες απαντήσεις να εξευρεθούν σε αυτά τα ερωτήματα γιατί διαφορετικά η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει μπούμεραν και θα μας χτυπήσει όλους πρέπει απόλυτα να αποσαφινιστεί τι γίνεται με αυτή την πρόταση της Επιτροπής και το, της διατάξης του ΠΟΕ και αν υπάρχει συμβατότητα ή όχι. Ιδίω όσον αφορά και την προστασία της υγεία που δεν καλύπτεται τώρα και σε σχέση με τις εθνικές διατάξεις που στο μέλλον θα ισχύουν, πώς μπορούν να διασφαλιστούν. Πρέπει να βρεθούν αυτές οι απαντήσεις τελικά και κατά πόσο, τα opt-outs, opting-outs, οι αυτοεξαιρέσεις είναι συμβατές ή όχι. Και τι σκέπτεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις διατάξεις ε, αυτές σε σχέση με τον ΠΟΕ. Τι θα γίνει, πώς θα τις προασπιστεί. Και από πλευράς Αυστρίας δημιουργείται και ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συνύπαρξη και τα δικαιώματα των διαφορετικών ε, χρηστών. Και εδώ σίγουρα σε σχέση με την παραγωγή στη Γεωργία που εμείς συμμετέχουμε, εμείς ως Αυστριακοί για την βιογεωργία και τα βιοτρόφιμα είμαστε, έχουμε ηγετικό ρόλο. Οι ισχύουσες διατάξεις δεν είναι προς ε, το συμφέρον μας με κανένα τρόπο. Και γι' αυτό το θεωρώ σημαντικό εμείς από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπομειστεί τις ευθύνες της και να μην τις απεμπολίσει. Και πολύ συγκεκριμένα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να έρθουμε σε επαφή και να δράσουμε συντονίζοντας τις απόψεις μας. Ευχαριστώ. Αν είμαστε γρήγοροι μπορούμε να δώσουμε στο λόγο στην Επιτροπή εντός του απογεύματος. Έχουμε άλλους πέντε εγγεγραμμένους να λάβουν τον λόγο. Θα είμαι σύντομη πρόεδρε. Και κατά τα άλλα επειδή θεωρώ σε σχέση με αυτό το θέμα η πρώτη προσέγγιση πρέπει να είναι θέμα αρχής και μετά θέμα ουσίας ε, και υπό αυτό το πρίσμα επίσης ε, από πλευρά του που παρουσίασε όλα τα περίπλοκα θέματα που δημιουργεί αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που εγώ απόλυτα συμμερίζομαι. Και αν τώρα το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι περίπλοκο και ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο και αν είναι επίμαχο και ξέρουμε ότι είναι επίμαχο, ε τότε πραγματικά δεν βλέπω πώς ενώπιον αυτής της περιπλοκότητας και του σύνθετου αυτού προβλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει απλά να θέσει τις ευθύνες στα κράτη-μέλη και εκείνη αποσύρεται και επιπλέον να θέσει τις ευθύνες και να επιβαρύνει τους ίδιους τους γεωργούς τους παραγωγούς. Όταν τα θέματα είναι δύσκολα, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, να περνάει η ευθύνη σε άλλους. Και όταν είναι εύκολα, τότε ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ρυθμίζει πράγματα και να εξομαλύνει ή να διευθύνει τις διαδικασίες. Μόνο που πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις ποιες είναι. Δεν, ε, δεν θέλω να επισέλθω τώρα στο θέμα της ουσίας, αλλά πώς είναι δυνατόν, πώς, τι θα κάνουν οι γεωργοί οι ίδιοι μέσα στην ίδια χώρα και πώς θα ανταγωνιστούν μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Μέχρι ποιου σημείου η παραγωγή, η παραδοσιακή παραγωγή και των βιολογικών προϊόντων δεν θα, επιζη... δεν θα ζημιωθούν με πρόσθετο κόστος όσον αφορά τις καλλιέργειές τους σε σχέση με τις γενετικά τροποποιημένες. Αυτό όμως σημαίνει να επισέλθουμε στα θέματα ουσίας και γι' αυτό περιορίζομαι εδώ. Πρέπει θέματα αρχής να εξετάσουμε και σε αυτό το επίπεδο πρέπει δυστυχώς να πω ότι αυτή η πρόταση δείχνει μια απευθυνοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απεμπόληση των ευθυνών της. Μια κατάσταση που νομίζω ότι πολιτικά ε, εξηγείται κυρίως. Λέγεται ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν θέματα περιβαλλοντικά ή της δημόσιας υγείας για να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Αυτή λοιπόν η απευθυνοποίηση, απεμπόληση ευθυνών είναι πολιτικό ε, μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα είναι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέμα. Όταν είναι περίπλοκα και σύνθετα τα θέματα και δύσκολα, φορτώνουν τις δυσκολίες σε άλλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό κάτι λέει. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς όλοι που οικοδομούμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δυνατόν μπροστά σε δυσκολίες, περίπλοκα θέματα και σύνθετα θέματα να απεμπολούμε τις ευθύνες μας. Η εικόνα που θα δοθεί σε άλλες χώρες με κάτι τέτοιο, για χώρες όπως η ΙΠΑ για παράδειγμα, θα πούνε ότι κανένας δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το γείτονά του. Δεν υπάρχει μια σταθερή, στεναρή θέση όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, όσον αφορά επιστημονικές θέσεις κοινωνικο-οικονομικές, περιβαλλοντικές και θέματα υγείας. Και όλα αυτά τους κάνουν να μην συμφωνούν και για να ολοκληρώσω, Πρέπει να δούμε διαφορετικά τα θέματα των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Πρέπει επιτέλους να επομιστούμε, να υιοθετήσουμε μια θέση που θα ξεκινά από θεμέλια επιστημονικά και έτσι να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό πρέπει υποχρεωτικά να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα περνάμε στον κύριο Σμιτ και μετά Πόλκα Νιέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάποια σχόλια προς τους συναδέλφους από τους πράσινους. Ε, ε, και εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Βλέπουμε αυτό, αυτή την πρόταση ως ε, ένα δούριο ύπο για την υπονόμευση της εθνικής ανεξαρτησίας για, που προσπαθεί να αχρηστεύσει κάθε κανόνες που βγαίνουν σε κρατικό ή και υποκρατικό επίπεδο. Ε, ο ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι να κατασταλάξει σε μια και αμετάβλητη άποψη ε, και ούτε πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα περνώντα τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με μια σωστή συζήτηση στη δική μας Επιτροπή, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλνιέτε και μετά Νίκολσον. Μάλιστα. Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί στη Λετωνία είναι ένα από τα θέματα που συζητιούνται πιο πολύ. Και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή δήμοι και κοινότητες που είναι επισήμως αναγνωρισμένες και αποτελούν το 75% της επικράτειας έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν γενετικώς τροποποιημένα. Και αυτό δείχνει σε τι βαθμό είναι απαραίτητο να το συζητήσουμε το θέμα. Τονίζω ότι όσο δεν θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια κοινή θέση επ' αυτού, και δεν θα δεσμεύεται βέβαια από τα μεγάλα μονοπόλια και τους μεγάλους παραγωγούς μέχρι τότε πρέπει οι χώρες να έχουν την ευθύνη για να παίρνουν τις αποφάσεις τους επί τέτοιων θεμάτων. Ευχαριστώ κυρία Καλινιέτε. James Nicholson και μετά θα κλείσει η Μαγκίνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι καλό που η εισηγητής μας είπε από την αρχή πολύ ρεαλιστικά πώς έχουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν φοβερές διαφωνίες και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε εύκολα να βρούμε μια λύση. Υπάρχει καμία δικαιολόγηση για την επανεθνικοποίηση αυτών των αποφάσεων, δεν ξέρω. Μερικοί λένε ότι γενικώ πρέπει να νομοθετούν περισσότερο τα κράτη-μέλη από ό,τι η Ένωση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ισχύει για 27 χώρες μέλη. Για μερικές θα ισχύει, για άλλες όχι. Και για να είμαστε, να πούμε και του στραβού το δίκαιο στραβός όνο επίτροπος, πρέπει να πούμε ότι μέχρι κάποιο βαθμό η αντίδραση του Συμβουλίου τον έπληξε και εκείνον. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πρώτα αν υπάρχουν εγκρίσεις, αν να ποιοι είναι υπέρ δηλαδή των γενικών τροποποιημένων. Δεν ξέρω. Αλλά αμφιβάλλω σοβαρά αν αυτό θα επιταχύνει τα πράγματα, η πρόταση δηλαδή της Κομισιόν. Ο εισηγητής έχει δίκιο, πρέπει να δοθεί μια νομική γνωμοδότηση για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Επίσης θα ήθελα να είναι σίγουρο ότι θα έχουν όλη επιλογή. Κόβω, κόβω πρόεδρε, δεν τα λέω όλα λοιπόν. Η Επιτροπή μας δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Αυτό αποκλείεται. Πρέπει να συμμετάσχουμε στην διαδικασία και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε μία λύση μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, James. Μαρία Βεγγίνες από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύναμη. Ευχαριστώ τον George Lyon που έθεσε πολύ λακωνικά τα ζητήματα για τα οποία θέλουμε απαντήσεις και θέλω πραγματικά να δω όλες αυτές τις νομικές γνωμοδοτήσεις, όλες αυτές τις νομικές γνώμες, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια δεν θα είμαι σκληρή απέναντι στην Κομισιόν, θα είμαι σκληρή απέναντι στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι πολιτικά τα μέλη του Συμβουλίου πραγματικά παρετήθηκαν του ζητήματος. Ε, καλό θα είναι να απαγορευτεί η εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών για τις ζωοτροφές μας, γιατί υπάρχει έντονος φόβος για τις γενετικά τροποποιημένες ουσίες. Έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ για το αν τα κράτη-μέλη θα έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν ή να περιορίζουν την καλλιέργεια. Δεν μιλούμε για την βούληση απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, τη διαδικασία ε, άδεια. Ε, είναι μια πολύ συγκεκριμένη και ειδική πρόταση. Για άλλη μια φορά, όπως είπε ο James Nicholson, θέλω πολύ να ακούσω τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ξέρω, George, αν θα έχεις χρόνο να πεις κάτι, ε, το να το απορρίψουμε θα μας, θα έρθουμε, το να απορρίψουμε αυτή την πρόταση θα μας φέρει προς τα πίσω. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ντόροθη Αντρέ έχει τον ε, λόγο και θα κλείσουμε αυτό τον πρώτο γύρο συζήτησης με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά παρόλα αυτά να θέσω και ορισμένα θέματα που έθεσαν οι βουλευτέ. Καταρχήν σας υπενθυμίζω ότι 13 χώρες μέλη ζήτησαν από την Κομισιόν τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2009 μάλλον, να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφασίζουν αν θα καλλιεργούν ή όχι γενετικώς τροποποιημένα. Και αυτό οφείλεται στο ότι τα πράγματα είναι παγωμένα στο Συμβούλιο ως προς τις αδειοδοτήσεις και η Κομισιόν με βάση επιστημονική γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ ζήτησε από τα κράτη-μέλη να αφαιρέσουν τη ρήτρα ασφαλείας. Επανειλημμένως όμως τα κράτη-μέλη σε επίπεδο Συμβουλίου δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχει θετική γνωμοδότηση ή άδεια της ΕΦΣΑ αλλά εμείς δεν αφαιρούμε τη ρήτρα ασφαλείας. Και η Κομισιόν ξανά έκανε επανειλημμένως τέτοιες προτάσεις και πάγωσαν τα πράγματα. Ο πρόεδρος Μπαρόσο λοιπόν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του δήλωσε ότι η Κομισιόν θα προτείνει κάτι, θα πρότεινε κάτι όπου θα δινόταν ενωσιακή αδειοδότηση με επιστημονικά στοιχεία αλλά θα είχαν την ελευθερία τα κράτη-μέλη να καλλιεργήσουν ή όχι. Τώρα βλέπω ότι όταν προσπαθεί ότι λέτε ότι η Κομισιόν προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της, όχι. Εμείς συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τις άδειες. Στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν με πλειοψηφία υπέρ κατά τις αδειοδοτήσεις για γενετικώς τροποποιημένα. Εμείς πάντα αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν τις αναλαμβάνουμε. Απλώς ακούσαμε το αίτημα 13 χωρών μελών. Λοιπόν, τώρα η πρόταση αυτή είναι ή όχι συμβατή με τον ΠΟΕ. Νομίζουμε ότι είναι συμβατή με τον ΠΟΕ. Γιατί είναι πρόταση που αφορά την καλλιέργεια και όχι την εμπορία σπόρων. Ζητιέται από τα κράτη-μέλη να σεβαστούν ορισμένα κριτήρια, το μέτρο αυτό δηλαδή να συμφωνεί με τη συνθήκη και με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Βάλαμε επίσης ως κριτήριο άρνησης το ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιστημονικά επιχειρήματα γιατί αυτά έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά την αποξιολόγηση και την αδειοδότηση Μόνο στα πλαίσια της ρήτρα ασφαλείας μπορούν να δεμαναλάβουν. Και είπαμε ότι είναι πέρα από τα επιστημονικά μπορούν να το επικαλεστούν. Και τώρα συζητούμε στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας, για τον ορισμό των κριτηρίων. Βεβαίως η Κομισιόν δεν είχε προτείνει συγκεκριμένο κατάλογο, ούτε πρόκειται να προτείνει κλειστό κατάλογο, πάντα ανοιχτό θα είναι, για να δίνεται πάντα η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιλέξουν και δεν πρόκειται να φτάσουμε στον καθορισμό όλων των κριτηρίων σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι βασικό να υπάρχει μια ελαστικότητα, ένα περιθώριο στα κράτη-μέλη, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να βελτιώσουμε αν χρειαστεί τα πράγματα και να δώσουμε στοιχεία που μπορεί να μην έχουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη τώρα σε περίπτωση που το μέτρο που θα λάβουν σε εθνικό επίπεδο είναι μεμπτή θα τύχουν προσφυγής. Νομίζουμε ότι οι αγρότες και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι του τομέα αυτού ίσως να ενδιαφερθούν περισσότερο στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να απαγορεύσει μια καλλιέργεια παρά από τις συζητήσεις στο επίπεδο της ΕΦΣΑ και για τη ρήτρα ασφαλείας. αν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει αρνητική επίπτωση στην αγορά, όχι, διότι σας είπα απαγορεύονται πιθανά μόνο καλλιέργειες και όχι και εμπορία των σπόρων και όλοι συμφωνούν ότι το θέμα αυτό δημιουργεί πολλές διαμάχες και δεν έχουμε καμία πρόθεση να το χρησιμοποιήσουμε ως προηγούμενο αν τώρα η Κομισιόν έκανε υπερβολικά νωρί τι προτάσει αυτέ πρόωρα και δεν έπρεπε να περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου. Εμείς την πρόταση αυτή την κάναμε σε συμφωνία με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008 που ζητούσε διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων τη λήψη υπόψη των, της περιφερειακής διάστασης και της συνύπαρξης των καλλιεργειών και υπάρχει ακριβώς το κείμενο αυτό της σύστασης για τη συνύπαρξη που προτείνει στα κράτη-μέλη να έχουν το δικαίωμα σε ορισμένες περιφέρειές τους να απαγορεύουν ή να μειώνουν την καλλιόργεια γενετικώς τροποποιημένων. Τι συζήτηση έγινε από το Συμβούλιο Γεώρ Περίβ, εδώ δεν ξέρω, είμαι απεσιόδοξη ε, υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά υπάρχουν και πολλά κράτη-μέλη που υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν και τη θεώρησαν θαραλέα. Και μάλιστα μας ζήτησαν να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα κριτήρια αναμένουν δε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Φυσικά αυτό που περιμένουμε είναι να μας πει ότι συμφωνεί, ότι δεν παραβιάζει τις αρχές ούτε τις συνθήκες ούτε του ΠΟΕ. Τα κράτη-μέλη δεν ζήτησαν από την υπηρεσία αυτή τη γνωμοδότηση, δεν ξέρουμε γιατί τη ζήτησαν, θα δοθεί σε λίγο. Θέλουν να την δουν πρώτα και μετά να επεξεργαστούν τα κριτήρια. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη πολλά βέβαια και είμαστε διατεθειμένοι να λύσουμε οποιαδήποτε τυχόν απορία να ξαναεξηγήσουμε την πρόταση και να σας βοηθήσουμε στην κατανόησή της. Νομίζουμε πάντως ότι πρόκειται για θετική πρόταση και που κανονικά θα βελτιώσει το υπάρχον σύστημα, διατηρεί δε την ενωσιακή αδειοδότηση με επιστημονικά δεδομένα και ενδυναμώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008, δηλαδή η αξιολόγηση του κινδύνου, ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Σε λίγο θα γράψουμε μία έκθεση με βάση στοιχεία από τα κράτη-μέλη για την κοινωνικονομική επίπτωση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και συνεχίζουμε να επιτηρούμε τη δραστηριότητα των μήκη όμικρων και των κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση του θέματος που μόλις εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν σε λίγο. Πολλά κάνουμε όπως βλέπετε, πολλά. Και, και θα καταλήξουμε σε όλα αυτά. Σύντομα και θα σας υποβάλουμε τα συμπαράσματά μας ας πούμε αυτή την έκθεση για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις τα τέλη του έτους. Προσπάθησα να είμαι σύντομη. Ορίστε. Ωραία. Ας ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας ευχηθούμε καλή τύχη στον George Lyon. Θα διατηρηθούμε σε στενή επαφή. Αύριο το πρωί. George, θε, Γιώργο, θες, να πάρεις το λόγο γιατί πρέπει να κλείσουμε πια. Ε, 20 δευτερόλεπτα. Μόνο ένα σημείο. Ο συνάδελφος ο Στεφάν Λεφόλ ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό μπορούμε να έχουμε κάποια, τυπικό διακανονισμό με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για αυτή τη νομική πρόταση. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δύο επιτροπές δεν μπορούν από κοινού να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα, να ασχοληθούν με ένα ζήτημα. Νομίζω πρέπει να δούμε αν μπορούμε να επισημοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Θα μας διευκολύνει πάρα πολύ να καταλήξουμε σε κάποιες συμπεράσματα, το να έχουμε κοινά, κάποια κοινή δουλειά. Εντάξει, Τζόρτζε, θα το φροντίσω, θα μιλήσω και μαζί σου και θα οργανώσουμε από κοινού τη διαχείριση αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Αύριο θα είμαστε στην αίθουσα 3C50. 3C50. Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι θα υπάρξουν δύο συναντήσεις. Μία στην ε, Βία Καμπεσίνα στον, στην αίθουσα των βουλευτών. Ξεκινάει τώρα και μια άλλη πρόσκληση από τον κύριο Ντανέλη για την ποιότητα των αγροτικών ε, προϊόντων στις 8.30 ώρα στην αίθουσα 5C2. Ευχαριστώ, θα τα πούμε αύριο. Συνάντηση των συντονιστών αύριο στις 9. Θα έχουμε πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Γεια σας.